Right, could everybody take their Παρακαλώ να καθίσετε όλοι. Σας δώσαμε ένα χρονικό περιθώριο. Έτσι για να, για να συνηθίσετε ότι έχουμε όλοι ξαναμπεί στο Λούκι. Καλή χρονιά σε όσους δεν μπόρεσα ακόμα να χαιρετήσω. Χρόνια πολλά. Και το πρώτο θέμα στην μέση η έγκριση. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 3η και 4η Μαου, τη 14η Ιουνίου, 23η Πρώτη, 22η Ιουνίου, 4η και 5η Οκτωβρίου, 8η και 9η Νοεμβρίου του 2010. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά, τα έχετε όλοι λάβει εντωμεταξύ πιστεύω. Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ουσία της ε, ακρόασης για την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την κύρια εισήγηση θα κάνει ο Επίτροπος Σέμετα. Μετά θα γίνει μια συζήτηση κοινή για να περάσουμε στη συνέχεια στις ε, παρουσιάσεις από το παρελθόν εμπειρονομών μας. Και άλλη κοινή συζήτηση στη συνέχεια. Μια και έχουμε λίγο καθυστερήσει, χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σέμετα τον οποίο είδαμε και πολύ πρόσφατα. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε που είχε την καλοσύνη να μας ξαναεπισκεφθεί. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και όλους όσους ε, δεν είχα την ευκαιρία να ε, ευχηθώ μέχρι τώρα. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας και την ε, Πρόεδρο για την πρόσκληση σε αυτή την συζήτηση για την κυριοτόμπο χρηματοπιστή για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότηση. Ύστερα από την πρόταση λοιπόν για νέα μέσα για την ενοποίηση των αγορών, τη σταθεροποίηση μάλλον των αγορών, την αντιμετώπιση των ε, χρηματοπιστωτικών διακυμάνσεων και την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. κατατίθενται προτάσει για το 2010 έτσι ώστε να περιγράψουμε στα θέματα αυτά. Με την ανάλυση στην οποία προβαίνουμε, καταλήγουμε στο συμπεράσμα ότι ορισμένα από τα ε, μέσα και για το μέρισμα και για τη λειτουργία των αγορών μπορούν να ενισχυθούν με την φορολόγηση του κινδύνου, του, της διακινδύνευσης μάλλον της αλλά και των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση της κυρίας Ποδηματά για, τη χρηματοδο... για την φορολόγηση των ευρω... για τα ευρωμόλογα, για τη χρηματοδότηση των πολιτικών συνελεχών και για τη χρηματοδότηση κλιματικής αλλαγή, μάλλον καλύτερα φο... τον φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω ότι εξή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι συμβάλλει κατά τρόπο υγιή και στέρεο στα δημοσιονομικά. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση στην συμπεριφορά της αγοράς στην υπόθεση αυτή, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει βεβαίως να ε, μην προβληθούν στην ενιαία αγορά λόγω της αγωγής των νέων φόρων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επιπλέον εμπόδια. Έτσι λοιπόν για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ανακοίνωση της, ε, του Οκτωβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα εξής. Ένας φόρος ε, για τις οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελεί μια καλή ε, λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, υφίσταται δίκαιη και ισότιμη φορολόγηση ως προς τα εισοδήματα και μπορεί να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό με περισσότερη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών μαζί με τη φορολόγηση και των μισθών αλλά και κυρίως των πριν που λαμβάνουν τα στελέχη. Ε, αυτό, άλλωστε το συνιστά και το Διεθνέ Ταμείο και στην πλειονότητά του ε, οι ειδικοί, επιστημονε, ε, πανεπιστημιακοί κύκλοι κτλ. Μια τέτοια πρόσοδος από ένα τέτοιο φόρο θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα πρέπει ένα τέτοιο μέσο βεβαίω να ενταχθεί με πολύ μεγάλη προσοχή στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και με ένα ποσοστό 5% θα μπορούσε να προσφέρει ποσοστά ε, μάλλον ποσά εσόδων 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη των 27, δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη των 27. Μια άλλη ανάλυση επίσης δείχνει ότι η επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα είναι πολύ χαμηλότερη με τον ειδικό αυτό φόρο των προσωπικών συναλλαγών και το περισσότερο βάρος θα τον αλάβει ο χρηματοπιστωτικό τομέα από την εισαγωγή αυτού του φόρου για την ανταγωνιστικότητα τώρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη να αναλύσει την ενδεχόμενη, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας τέτοιος φόρος στην εισαγωγή. Ε, έτσι ώστε να υπολογιστεί και το κόστο που μπορεί να προκληθεί για του χρηματοπιστωτικού μα οργανισμού. Ο κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα πάντω, από ό,τι υπολογίζεται θα είναι πολύ χαμηλότερο από την εισαγωγή ενό τέτοιου φόρου από ότι ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, που προτείνεται. Συνολικά και σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ανάλυση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την προαγωγή μιας συμφωνίας με τους πιο σημαντικούς οικονομικούς εταίρους. Εγώ προσωπικώς έθεσα το ζήτημα και με το Υπουργείο των Οικονομικών των ΗΠΑ το Δεκέμβριο και διαπίστωσα καλή διάθεση εκ μέρου των Αμερικανών ομολόγων. Ε, όταν δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη δική μα αξιολόγηση επιπτώσεων, είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν και πάλι μαζί μα. Δεδομένου ε, του υψηλού, των υψηλών εισόδων που μπορεί να προκαλέσει αυτός ο, να, να γεννήσει μάλλον αυτός ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα ποσοστό 0,1% που θα σημαίνει 60 δισεκατομμύρια ε, ευρώ έσοδα. Υπάρχουν ακόμη εκτιμήσεις δεκαπλάσιων εσόδων από ορισμένες μελέτες, οι οποίες υπολογίζουν και τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Αλλά αυτές τις εκτιμήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θεωρεί μάλλον αβέβαιες. Έως το 2011 λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μια μελέτη επιπτώσεων και με την αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτών των ε, ρυθμίσεων των ε, τελών για τις τράπεζες και των σχετικών φόρων. Πού έχουμε φτάσει τώρα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουν, γίνει μελέτες, έχουν ξεκινήσει μάλλον οι μελέτες ε, για τον ε, φόρο που θα επιβαρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη σχετική τιμολόγηση και τις αντιδράσεις των αγορών σε μια νέα φορολογία και το κίνδυνο να χαθούν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα μετακινηθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεσεις με εξωτερικούς ε, οργανισμούς ή φορείς, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Διεθνών, ε, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ε, και, άλλες, και άλλοι διεθνείς φορείς όπως και πανεπιστημιακοί έχουν ήδη αρχίσει να εμπλέκονται σε αυτή τη μελέτη για να δούμε και με πρότυπα το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Προσπαθούμε δηλαδή με πρότυπα να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις και στο κόστος του κεφαλαίου και στην ανάπτυξη και στον, στην ανάληψη κινδύνου. Για να αξιολογήσουμε περισσότερο λοιπόν τα σωρευτικά μέσα, οι διάφορε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναπτύξει πολύ στενή συνεργασία ω προ τι επιλογέ που αναλύονται. Θα εκτιμηθεί το κόστο ενό ε, φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, μόνο για την Ευρώπη, καθώς και ο κίνδυνος μετακίνησης ε, των επιχειρήσεων. Και βεβαίως θα δούμε και σε σχέση ε, με τον ε, φόρο ε, κεφαλαίων, επί των κεφαλαίων, τι είδου επιπτώσει μπορεί να έχει και σε τι ποσοστά μπορούμε να τον ορίσουμε. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κατάλληλε προτάσει και πρωτοβουλίε για την σωστή φορολόγηση συγγνώμη, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω στο επόμενο θέμα που ε, εγείρει η έκθεση τη κυρία Ποδηματά και που είναι η φορολογία του άνθρακα, του οξυδίου του άνθρακα. Καταρχά, θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχαρίστησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη την οποία εκφράσατε ω προ την οδηγία, ω προ την θέσπιση μια οδηγία για φορολόγηση του οξυδίου του άνθρακα δηλαδή φορολογία ουσιαστικά των ενεργειακών προϊόντων. Ε, αυτή η φορολόγηση μπορεί να έχει δύο κυρίου στόχου. Πρώτο, να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα έξω από το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγή εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Και δεύτερον, να εξορθολογήσει αυτήν την φορολόγηση συνδέοντας την με το ενεργειακό περιεχόμενο έτσι ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις που προέρχονται από διαφορετικές ενεργειακές πηγές. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί τώρα στην, ε, στην μελέτη επιπτώσεων καθώς και στην αναθεώρηση των υφισταμένων οδηγιών και πρόκειται πολύ σύντομα να καταθέσω την επίσημη πρόταση έτσι ώστε να έχουμε μια γερή βάση για συζήτηση με τα κράτη-μέλη στο σημαντικό αυτό θέμα. Διαβλέπω επίσης οικονομικές ευκαιρίες ως προς την αναθεώρηση του συστήματος των εκπομπών, όπου πιστεύουμε ότι μπορεί μια πράσινη φορολογία να ενθαρρύνει και την, πράσινη καινοτομία, και την ενεργειακή καινοτομία και η αναθεώρηση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για την αναδιάρθρωση των φορολογικών συστημάτων από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να αναπτυχθούν συστήματα φορολογικά τα οποία θα αποτελούν και κίνητρα για την ανάπτυξη νέων συνεργασία και πράσινων ενεργειών. Και βέβαια θέλουμε να αποφύγουμε τη φορολόγηση ε, του εργατικού δυναμικού, του, της εργασίας δηλαδή, που θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Ξέρω ότι έχετε συζητήσει και την δυνατότητα της ε, προσαρμογής των ε, φορών η κατανομή των αδειών και διανομή αδειών ε, σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν ε, ένα καλό κίνητρο για την αποφυγή των ε, εγκρών διοξιδίου του άνθρακα. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια μελέτη της διαπιστώνει ότι τα μέτρα αυτά ήδη επαρκούν στις ισχύουσες συνθήκες. Πλην όμως συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τον κίνδυνο του διοξιδίου του άνθρακα και να αναζητούμε ισοδύναμα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Η έκθεση κυρία Ποδηματά επίση αναφέρεται στην ιδέα της αγωγή ενό φόρου προσθέμενης αξίας διοξιδίου του άνθρακα έτσι ώστε να συνδεθεί το ε, θέμα των νεκρών διοξιδίου του άνθρακα με την εσωτερική παραγωγή. Αυτή την ε, πρόταση όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την εξέτασε περαιτέρω, διότι θα συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο σύστημα. Επιπλέον, ένας φόρος τύπου ε, προσθέμενης αξίας έχει το μειονέκτημα ότι ο τελικός ιδιώτης καταναλωτής είναι εκείνος ο οποίος επιβαρύνεται με τον φόρο αυτό και ως εκ τούτου ε, δέχεται και να προκαλέσει αλλαγές συμπεριφοράς σε ολόκληρη την καταναλωτική αλυσίδα. Ανεπιθύμητες αλλαγές. Και τώρα θα ήθελα, Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να προχωρήσω για τα ευρωομόλογα με ορισμένε σύντομε ε, παρατηρήσεις για να είμαι πιο σαφή ω προ τα ευρωομόλογα. Δεν θα, ε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν αναφέρομαι στι δηλώσει του Προέδρου Μπαρόσο ω προ την κατάσταση τη Ένωση και δι αυτέ τι δηλώσει που προβλέπουν θέσπιση ομολόγων για τη χρηματοδότηση μεγάλων ε, σχεδίων υποδομών, των ομολόγων σχεδίων δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με την ε, προσέλκυση χρηματοδότησης ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άλλους οργανισμούς και την ιδιωτική κεφαλαία αγορά. Τουναντίον, θα ήθελα να αναφερθώ στα ευρωομόλογα ως ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης ή μάλλον διαχείρισης χρέους, ε, το οποίο θα καλύπτει μέρος του κρατικού χρέους. Έχουμε εδώ να κάνουμε, του δημόσιου χρέους καλύτερα, έχουμε να κάνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά όμως τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν Προ το παρόν δεν φαίνεται να είναι όριμη η περίοδος για να συζητηθεί το θέμα αυτό απευθείας. Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητα και τον σχετικό μηχανισμό που επιτρέπουν ε, τον δανεισμό για τα κράτη-μέλη τη ζώνης του ευρώ μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνούς Ταμείου. Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2010, ε, οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός μέσου διαχείρισης κρίσεως προχωρούν και θα καταλήξουν σε αποτελέσματα κάποια στιγμή. Και είμαι βέβαιο ότι οι συζητήσει σημερινέ θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή ω προ την ιδέα μια καινοτόμου χρηματοδότηση, την αναζήτηση μια καινοτόμου χρηματοδότηση. Μπορούμε, νομίζω, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση αυτή τη σε αυτού του τομέα και βεβαίως οι υπηρεγνώμονε τη υπηρεσία μου είναι στη θέσή σα για να σας στηρίξουν και εσάς και τα μέλη του πάνελ και προσβλέπω σε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ, Σας Ήσασταν συντομότατο και σας ευχαριστούμε. Μπορέσαμε να καλύψουμε ένα μέρος της καθυστέρησής μας, γιατί αργοπορήσαμε στην αρχή της συνεδρίασης. Η κυρία Ποδηματά έχει ζητήσει τον λόγο, Άννη. Uh, Ευχαριστώ Σάρων, αγαπητέ Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχηθώ στην Ομίγυρη. Καλή και ευμερούσα χρονιά. Τώρα θα μιλήσω στα ελληνικά, επιτρέψτε μου, Επίτροπε. Ερωτήματα με τη σειρά που τοποθετηθήκατε κι εσείς, πρώτα απ' όλα σε σχέση με, την, ε, με το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσής μου για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα το φόρο άνθρακα και τέλος τη συζήτηση για τα, για τα ευρωομόλογα. Σε ό,τι αφορά την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ε, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων εδώ με τους στόχους που περιγράψατε, ε, ότι θέλετε ε, να υπηρετήσετε προχωρώντας ένα τέτοιο μέτρο. Και αναφερθήκατε σε τρεις ε, συγκεκριμένες κατηγορίες. Είπατε ότι θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συμβάλλει με δίκαιο και ουσιώδη τρόπο στα έσοδα. Το δεύτερο σημείο που υπογραμμίσατε ήταν ε, η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα να συμπληρώσει το νέο πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αναφερθήκατε μάλιστα και το συγκράτησα αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο double dividend, στο διπλό όφελος δηλαδή που προκύπτει από τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, χωρί φυσικά όλοι επίση το συμμεριζόμαστε αυτό να δημιουργηθούν προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, και το τρίτο, ε, να μην δημιουργηθούν επιπρόσθετα εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ε, η ερώτησή μου, κύριε Επίτροπε, είναι ακριβώς σε ό,τι αφορά το δεύτερο κριτήριο που υπογραμμίσατε. Την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ως συμπληρωματικού εργαλείου για την καλύτερη ρύθμιση και ε, εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και θέλω να σας ρωτήσω, ε, ο φόρος, ο φόρος επί των κερδών, το Financial Activity Tax που είναι πολύ καθαρό και από τη σημερινή σας παρέμβαση ότι τον προκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το ότι θα μου επιτρέψετε να πω ασφαλώς ε, το ίδιο εισηγείται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά στο επίπεδο το ευρωπαϊκό δεν έχουμε ακόμη. Θα έχουμε το καλοκαίρι, όπως είπατε και εσείς, μια πλήρη και ενδελεχή μελέτη επιπτώσεων για το ποια είναι η καλύτερη επιλογή με βάση αυτά τα τρία κριτήρια που μόνο σας ε, αναφέρατε και τα οποία συμμεριζόμαστε. Ε, ο φόρος λοιπόν επί των κερδών, το Financial Activity Tax, είναι σαφές νομίζω ότι δεν υπηρετεί αυτό το δεύτερο κριτήριο που έχει για μας ιδιαίτερη σημασία, το να λειτουργήσει δηλαδή η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ως συμπληρωματικό εργαλείο για την καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλώς. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων. Ε, το, το θέμα μας είναι με ποιο τρόπο θα είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει και να ασκήσει πίεση στο παγκόσμιο επίπεδο, στο επίπεδο του G20, προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, άρα λοιπόν το ερώτημά μου εστιάζεται σε αυτό, ε, στον double dividend και στον, ε, στον ρόλο που πρέπει να έχει φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ως συμπληρωματικού εργαλείου για την καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και βεβαίως μιλήσατε για τη μελέτη επιπτώσεων αλλά πάλι έχουμε την εντύπωση ε, σαν να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προαποφασίσει ποια είναι η καλύτερη επιλογή, ε, χωρίς ε, να έχει γίνει αυτή η λεπτομερής μελέτη επιπτώσεων. Σε σχέση με την φορολόγηση του άνθρακα, νομίζω ότι συγκλίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, συμμεριζόμαστε τα κριτήρια που βάζετε, υποστηρίζουμε την αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, ε, φορολόγηση της, ε, της ενέργειας με τα κριτήρια που θέσετε. Και το τρίτο, για να μην μακρηγορώ, σε σχέση με τα ευρωομόλογα, κύριε Πίτροπε, αφήνω και εγώ με τη σειρά μου στην άκρη τα ευρωομόλογα σύμφωνα ως εργαλείο αναπτυξιακό χρηματοδότησης μεγάλων ευρωπαϊκών σχεδίων, μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών, έργων υποδομών και έρχομαι στη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ευρώπη ε, σε μια σειρά ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στα ευρωπαϊκά όργανα, για τα ε, ευρωομόλογα ε, ως εργαλείου διαχείρισης τμήματος του δημοσίου χρέους. Και είπατε, κύριε Επίτροπε, ότι δεν είναι η στιγμή για να γίνει αυτή η συζήτηση. Και εγώ αντιθέτως έχω την εντύπωση ότι ακριβώς τώρα είναι η στιγμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι αυτό δεν προκύπτει μόνο από τη δική μου δήλωση, προκύπτει από μια σειρά πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που έχουν έχουν ε, ε, παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, το κοινό άρθρο ε, του Προέδρου του Eurogroup, του κυρίου Juncker και του κυρίου Τρεμόντι στους Financial Times, πρωτοβουλίες από think tanks, από οικονομολόγους. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε όλη την ίδια γνώμη, αλλά θέλω να επιμείνω στο σημείο που είπατε ότι δεν είναι η στιγμή να το συζητήσουμε. Πώς είναι δυνατόν όταν η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αυτές τις διαστάσεις όλο το τελευταίο διάστημα, όταν αποδεδειγμένα οι απαντήσεις και ε, οι λύσεις τις οποίες έχουμε κατευθυνθεί μέχρι σήμερα αποδεικνύονται ανεπαρκείς να απορρίπτουμε χωρίς να εξετάσουμε σε βάθος μια τέτοια πρόταση. Και θέλω με την ευκαιρία να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τελευταίο ψήφισμα που υιοθέτησε με πρωτοβουλία της δικής μας Επιτροπής για τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσης ε, λίγο πριν, μια μέρα πριν συγκληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου σαφώς ζητάει από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει αμέσως σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει σε μια ενδελεχή ε, μελέτη ε, σε σχέση με αυτήν την, επιλογή, την έκδοση ευρωομολόγων ως εργαλείου διαχείρισης τμήματος του δημοσίου χρέους και ως μια ευρωπαϊκή απάντηση, μία από τις ευρωπαϊκές απαντήσεις που θα μπορούσαν να πείσουν τις αγορές στην διευρυνόμενη ε, κρίση που ε, υπάρχει σήμερα στην ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank um, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εφόσον είναι η συγγήτρια η Άννη, είναι λογικό να μακρηγορεί σε σχέση με άλλα μέλη της Επιτροπής. Και θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσως στον Επίτροπο για να ακούσουμε τις απαντήσεις του και προς το παρόν έχουμε Φέγγι Γκόλντ και τη Σίλβι Γκουλέρτ ε, στον κατάλογο των ομιλητών και εσάς βεβαίω, ναι. Ένα λεπτό και θα σας σημειώσουμε όλους τον κατάλογο. Ε, στο μεταξύ ας ακούσουμε τον Επίτροπο. Ε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά. Ελπίζω να είναι παραγωγική. αληθεύει ότι μας περιμένει σκληρή δουλειά αυτή τη χρονιά ε, στους τομείς αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας κυρίως. Ως προς τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας τώρα για τον φόρο επί των κερδών, το FAT, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αναλύουμε το θέμα αυτού του φόρου επί των κερδών και επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, προτείνουμε και αναλύουμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις και για τα δύο είδη φόρων. Για το φόρο επί των κερδών, πώς τίθεται το δίλημα, αν θα χρησιμοποιήσουμε ευρεία ή στενή φορολογική βάση. Ε, για το φόρο επί των κερδών ε, επίσης αναλύσαμε τρεις εναλλακτικές λύσεις. on how the... Ανεξάρτητα από το πώς θα διαμορφωθεί, θα σχηματιστεί ο φόρος ε, επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, υπάρχει και το ενδεχόμενο να πραγματευτούμε και το θέμα του δεύτερου στόχου των εργασιών μας, δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε ως βάση τις ε, δραστηριότητες ανάληψης κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε το φόρο ούτως ώστε η ε, επικίνδυνη συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να φορολογείται, αυτό μας επιτρέπει να καλύψουμε και το δεύτερο στόχο, στον οποίο εσείς αναφερθήκατε. Ε, πλην όμως σήμερα είναι πρόωρο, κατά τη γνώμη μου, να αναλάβουμε ήδη δέσμευση σχετικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο ε, σχεδίασης του φόρου. Χρειάζεται ενδελεχής αξιολόγηση επιπτώσεων, πρωτήτερα, όπως ανέφερα και στην αρχική μου παρουσίαση, εργάζεται πολύ σκληρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Ε, με ρωτήσατε πώς τοποθετούμε και αναφερθήκατε στη στη θέση που ε, λαμβάνω. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στη, στη γνωμοδότησή σας, όπου όπου φαίνεται να έχει οθετήσει μια συγκεκριμένη στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση. Κοιτάξτε. Έχουμε ήδη εξαγάγει μια ανάλυση τον Οκτώβρη συγκεκριμένα το 2010 και επί τη βάση της ανάλυσης αυτής και των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας τότε, αναπτύξαμε και τον πολιτικό μας προσανατολισμό. Όμως αυτό δεν ε, σημαίνει ότι δεν θα διεξαχθεί ε, αξιολόγηση επιπτώσεων και όπως ήδη ανέφερα θα αναλύσουμε την αξιολόγηση, θα ε, προβούμε στην αξιολόγηση αντικτύπου για τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια ως προς το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενδελεχής αξιολόγηση αντικτύπου είναι μια εκ των όνου προϋπόθεση για τη συνέχεια. Όταν οριμάσει το θέμα, σύν το χρόνο, θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης αντικτύπου. Ε, τώρα διεξάγεται εξάλλου η αξιολόγηση αυτή. Οψόμεθα. Για τα ευρωομόλογα ε, είναι λίγα σημαντικό να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει σαφέστατες ε, δεσμεύσεις και θα κάνουμε εισηγήσει ε, σχετικά με την ανάπτυξη ε, μελλοντικών μηχανισμών. Δεν είναι θέμα του χαρτοφυλακίου μου τα ευρωομόλογα. Ο Επίτροπος Όλη Ρέν είναι αρμόδιος. Στο παρόν στάδιο πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μελέτη για τα ευρωομόλογα δεδομένης της ε, κρίσης ε, για το δημόσιο χρέος, για το πώς θα αντιδράσουμε σε συνολικό επίπεδο στην ε, κρίση και θα αναμένονται λίγαν συντόμως πολύ συγκεκριμένε προτάσεις από πλευρά της Επιτροπής. Πρόεδρος, τώρα έχουμε τέσσερα λεπτά και 9 ομιλητές. πιστεύω ότι μπορούμε αργότερα να κερδίσουμε λίγο χρόνο, συγγνώμη, αλλά θα ήθελα παρακαλώ να μιλήσετε για ένα λεπτό. Σφέν Σίλβιου, Ούντο, Λιπέρ Βάνς, Τόμας Μαν, Λενάρντο και Λάρς. Νομίζω τους είπα όλους. Το Λάρς, ο κύριος Μπουκρός. Σφέν Σίλβιου, Ούντο και Όλε. Πριν να ξανακούσουμε τον Επίτροπο. Και ας βάλετε και το χρονόμετρο, σας παρακαλώ, ένα λεπτό έκαστος. Μετά τις διακοπέ των Χριστουγέννων και μετά όλε τι λειτουργίε στην Εκκλησία ήλπιζα ότι η συζήτηση για τον των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα έπαιρνε μια κάποια όθηση σε χώρε όπω η Τινησία και η Αλγερία, οι οποίε αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση στι τιμέ των τροφίμων και που φαίνεται ότι χρειάζεται να ε, επιδείξουν ε, σοβαρότητα και στις υποσχέσεις τους. Πάντως φαίνεται ότι δεν ε, εμπνεύστηκε από το πνεύμα των Χριστουγέννων η Επιτροπή στην υπόθεση αυτή. Α συνεχίσουμε όμω την προσπάθειά μα. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, όχι μόνο τις επιλογές να εξετάζουμε, αλλά και το κόστος, όχι μόνο το πώς, αλλά και το τι θα χρεώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην παγκόσμια οικονομία, έτσι ώστε να έχουμε έναν πύχη, ένα ε, μέτρο σύγκριση. Τα 25 δισεκατομμύρια είναι πολύ λίγα σε σχέση με το εξωτερικό κόστος που προξενεί για την υπόλοιπη οικονομία ο χρηματοπιστωτικό κλάδος. Και γι' αυτό ελπίζω να συμπεριληφθεί και αυτή η ανάλυση. Επίση, καλώ ορίζουμε τι εργασίε σα ω προ το διοξείδιο του άνθρακα, ω προ τα ομόλογα για σχέδια ε, για υλοποίηση σχεδίων. Τα ευρωομόλογα όμως έχουν κρίσιμη σημασία και σκοπεύουμε να ζητήσουμε να συζητηθούν στο πλαίσιο αυτό με τον Όλυ Ρέν και σε μια περαιτέρω ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και για το ότι κάνετε στους ε, διάφορους τομείς με ιδιαίτερο κουράγιο. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω όμως ε, λίγο παραπάνω. Γιατί πραγματικά, ειλικρινά, υπάρχει κάτι το οποίο με θλίβει σε αυτά τα οποία λέτε. Η Κομισιόν έχει το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας για να έχει κανείς πρωτοβουλία θα πρέπει να προτρέχει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά ε, για την επαναχρηματοδότηση του χρέους ε, γιατί πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά και να ξέρουμε γιατί μιλάνε και εγώ ως εισηγήτρια για την ε, οικονομική διαχείριση το έχω πάλι στο κείμενο σχετικά με τις κυρώσεις για έναν απλό λόγο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι εκτός. Θα ήταν πραγματικά περίεργο να μιλάνε όλες οι εφημερίδες. Ο πρόεδρος του Eurogroup ε, να γράφει στο Financial Times ή μέσω της Zeit να απευθύνεται στην κυρία Μέρκελ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην έχει ιδέα για όλα αυτά. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε το Συμβούλιο να το σμπρώξει το θέμα ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε πραγματικά στην πρωτοπορία. Αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Η Γιούτα. Äh, Ο κύριος Τόμας Μαν. Ο κύριος Μπούρμαν, συγγνώμη. Πρόεδρε, θα ήθελα να δω μια στάθμιση μεταξύ των δύο φόρων των, του φόρου κεφαλαιοαγοράς και του φόρου επί των κερδών. Στο φόρο επί των κερδών λέτε κι εσείς ότι σημαντικός παράγον είναι η χρηματοδότηση και του ποσού των μισθών ή πριμ των χρηματοπιστωτικών ε, οργανισμών. Στον δε φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα είχαμε ως πλεονέκτημα ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν το high frequency trading θα φορολογούνται. Αλλά μας λέτε ότι αυτό είναι κακό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω τώρα εγώ. Γιατί. Και πώς διασφαλίζουμε ότι θα μείνουν επιχειρήσεις μέσα στην Ευρώπη εάν έχουμε φορολόγηση για τους μεγάλους ιδιώτες ε, ε, με τις πολλές θηγατρικές που παρέχουν συμβουλές στον ιδιώτη και παρέχουν ε, δάνεια για τον καταναλωτή και αυτό θα είναι ε, χρήσιμο να τους φορολογήσουμε, καλό. Αλλά εάν θέλουμε να ε, φορολογήσουμε εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν το μεγάλο κίνδυνο, μπορεί να αποσταθεροποιήσουν την αγορά και στη τελευταία ανάλυση κερδίζουν πάρα πολλά από αυτό το κίνδυνο, Μα λέτε ότι είναι κακό να του φορολογήσουμε. Εξηγήστε μου παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο να παρακολουθήσω το συλλογικό σα. Δεν μπορώ να σα καταλάβω. Όλε. Όλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Στα αλήθεια, νομίζω πως πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της φορολόγησης, αυτού του νέου συστήματος φορολογίας. Θα είναι ε, διατηρήσιμη, βιώσιμη φορολογική βάση ε, για το, τους φόρους του άνθρακα. Θέλουμε να είναι ευθύνουσα η πορεία ε, συν το χρόνο, έτσι, αλλιώς θα ήταν παράξενο. Και επίσης δεν πρέπει να παρεμποδίσει η λειτουργία της αγοράς. Και όλες αυτές οι δοκιμές για την αποτελεσματικότητα να τις κάνετε βεβαίως, αλλά ε, επειδή είστε ο ειδικό ε, στην Ευρώπη για τους φόρους, ε, καλό θα ήταν να μας πείτε εσείς ποιο από τα μέτρα θα προτιμούσατε, ιεραρχήστε τα κατά σειρά προτεραιότητας. Ίσως θα βοηθούσατε λίγο τη συζήτηση, τουλάχιστον στην Επιτροπή μας, κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ακούσω την άποψή σα. Εσείς τι προτιμάτε, ε, φόρο επί των κερδών, επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή όλο το πακέτο. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι συμπληρωματικοί φόροι θα λύσουν το πρόβλημα της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση. Θέλω να ακούσω και τη δική σα την άποψη, ο επίτροπο. Μάλλον καλό είναι να αρχίσω από το τέλος, από το τελευταίο ερώτημα. Πρώτον, ε, η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και η φορολόγηση του άνθρακα είναι δύο διαφορετικά είδη φόρων και σχεδιάζονται για να καλύψουν διαφορετικούς στόχους. Για την φορολόγηση των εκπομπών του άνθρακα, ο στόχος μας είναι να αναδιαρθρώσουμε ε, τον υφιστάμενο φόρο για τους ενεργειακούς πόρους τον εφιστάμενο άμεσο φόρο για τους ενεργειακούς πόρους, ούτω ώστε να τον προσανατολίσουμε προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και έτσι να άρουμε τα, τους φραγμούς για την εύρεθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αναδιάρθρωση λοιπόν του φόρου, αυτός είναι ο στόχος, για να δημιουργήσουμε φορολογικά κίνητρα και να είμαστε ενεργειακώς πώς αποτελεσματικοί, λαμβάνοντας ε, υπόψη τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής, να εξετάσουμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε όργανα μέσα της αγοράς για να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή μας αποτελεσματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η σωστή ρότα την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, ολοκληρώνουμε σταδιακά τις εργασίες μας ε, και ε, ταχύτατα θα υποβάλουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ας περάσω τώρα στην φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η προσωπική μου άποψη είναι η εξή. Είναι σαφή τα πράγματα κατ' εμέ από φορολογικής πλευράς. Όλοι γνωρίζουμε πως ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξαιρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον ΦΠΑ και Ένα από τα μέτρα που θα εισηγηθούμε για να αντισταθμίσουμε αυτό το χάσμα, επειδή δεν υπάρχει αυτός ο φόρος στο χρηματοπιστωτικό τομέα, έγκυται στο εξή. Επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε αναλύσει μέχρι τούδε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προτιμητέα λύση ήταν ακριβώς ο φόρος ε, επί των κερδών. Αυτό σαφέστατα ε, το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας προκρίνουμε αυτή τη λύση. Πριν όμως ε, λάβουμε την τελεσίδικη απόφαση και προτείνουμε συγκεκριμένα νομοθετήματα στον τομέα αυτό, θα πρέπει εις βάθος να αναλύσουμε όλες τις αναλλακτικέ λύσεις συμπεριλαμβανομένων ε, και των προτάσεων ε, για τους φόρους, παραδείγματος χάρη επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει των πληροφοριών που έχουμε και εμείς, αλλά και βάσει των μελετών που έχουν γίνει, μια αυστριακή μελέτη μεταξύ άλλων που κατά πάσα πιθανότητα θα συζητήσετε στην ακρόασή σας αργότερα, θέτει σοβαρότατα ζητήματα για ενδεχόμενη μετεγκατάσταση, μετατόπιση των χρηματοπιστωτικών συναλλάγων. Αυτό είναι ουσιαστικό και σοβαρό θέμα και οφείλουμε να το εξετάσουμε διεξοδικότητα για να προσαρμόσουμε, να διαμορφώσουμε εμεί το μέτρο του δυνατού τη συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι δυσχερέστατο αυτό το έργο και από αυτού εργάζονται οι, ε, οι υπηρεσίες μας. Ας περιμένουμε λοιπόν το πόρισμα τη ανάλυσή του και θα ε, υποβάλουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις όπως προείπα στον τομέα αυτό. Ε, τώρα, αν είμαστε προτεργάτες ή ουραγοί για τα φορολογικά θέματα, στην Επιτροπή εννοώ, ε, αντιλαμβάνεστε πως σχεδόν σε όλα τα βασικά έγγραφα και ανακοινώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνουμε ρήτρε και διατάξει για τα φορολογικά ζητήματα. Προχωρούμε με βήμα ταχύ στο τομέα της φορολογίας. Ποιο είναι το θέμα βεβαίως οι αποφάσεις επί των φορολογικών δεν μπορούν να αναλυφθούν ε, μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι περίπλοκα, πολύ σύνθετα ε, τα προβλήματα και αγγίζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Οφείλουμε να σπεύσουμε βραδέως, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, στις αναλύσεις μας. Στην αρχή της θητείας μου είχα αναφερθεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις στις διάφορες προτάσεις που τώρα επεξεργάζονται ε, ε, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημειώνεται ταχεία πρόοδος. Νομίζω ότι εν συντομία απάντησα. Ε, μήπως θα μπορούσατε να σχολιάσετε την ερώτηση του κυρίου Μπούλμαν, επίτροπε, μάλιστα. Ε, ο κύριος Μπούλμαν ρώτησε πώς, μάλλον κύριε Μπούλμαν, να τα ξαναπώ, Πρόεδρε. Η στάθμιση του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και επί των κερδών. Πώς του συγκρίνεται. Μας λέτε ότι ο φόρος επί των κερδών ε, θα επιβρυνθεί ως προς την, ε, τους μισθούς και τα κέρδη των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό να αποτελέσει μία λύση όταν αυτοί οι οργανισμοί προσφέρουν χρηματοδότηση, δάνεια κτλ. για τον ιδιώτη καταναλωτή και γιατί είναι κακό το να επιβαρυνθεί με ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο συναλλασσόμενος εκείνος, ο μεγάλος συναλλασσόμενος, ο οποίος επενδύει στον κίνδυνο και κερδίζει από αυτόν. Δεν μου φαίνεται πολύ, πιθανό, πολύ λογικό το επιχείρημά σας και γι' αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσετε περισσότερο. Ε, για αυτά τα δύο είδη φόρων, ε, κοιτάξτε, όπως σας είπα, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, των, επί κερδών, συγγνώμη, προσωμιάζει στον ΦΠΑ και άρα θα καλύψει αυτό το κενό της απουσίας του ΦΠΑ στον χρηματοπιστωτικό τομέα καλύπτοντας λοιπόν ε, τις ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το θέμα βέβαια είναι να τον διαμορφώσουμε, να τον σχεδιάσουμε αυτό το φόρο με τρόπο ώστε να μην μετακυλιστεί στους ε, καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τον ΦΠΑ. Εκείνοι ε, ε, υφίστανται το άχθος αυτών αυτού του φόρου. Επ' αυτού λοιπόν εργαζόμαστε και ε, διαρευνούμε τις πιθανές λύσεις. Ε, ως προς το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, ε, οι ακαδημαϊκές μελέτες ε, και διάφορες, ε, διάφορα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν καταλήγουν σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου θα μειώσει την αστάθεια των αγορών. Το αντίθετο δείχνουν μάλλον. Αυτές οι μελέτες καταλήγουν στο πόρισμα ότι θα αυξαθεί η νευρικότητα και η αστάθεια των αγορών. Με τις δύο προτάσεις, ε, ούτως ή άλλως πρέπει να προσέξουμε. Χρειαζόμαστε διεξοδική ανάλυση, να δούμε ποιος θα είναι ο πραγματικός, ουσιαστικός αντίκτυπος, αν ακολουθηθεί αυτή η εναλλακτική λύση. Για το θέμα του ποιος θα καταβάλει αυτό το φόρο σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης μας, ε, καταδεικνύεται ότι είναι πολύ ευκολότερο να υποστεί ο καταναλωτής ε, το φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε σχέση δηλαδή με το φόρο επί των κερδών, γιατί οι συναλλαγές για τους καταναλωτές ε, γίνονται και οι φορείς ε, της χρηματοπιστωτικής αγοράς εύκολα στην τιμή τους μπορούν να καλύψουν, να μετακυλήσουν στο λογαριασμό που πληρώνει ο καταναλωτής το φόρο αυτό. Οπότε θα πρέπει να εισηγηθούμε και εναλλακτικέ ε, λύσει να μελετήσουμε το θέμα και να ε, διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτό τον φορό ώστε να μην υπάρξει αυτή η μετακύληση της τιμής ε, στον καταναλωτή. Μάλιστα τώρα είμαστε σε απόγνωση, δεν έχουμε καθόλου χρόνο στη διάθεσή μας, λέει η πρόεδρο, η Περβάνς Περές, Ντανίτα Χιούμπνερ, Τόμα Μαν, Λεωνάρντο, Ντομινίκ και η κυρία Κρός ε, στη συνέχεια. Περβάνς, μήπως έχεις δηλώσεις και όχι ερωτήσεις. Euh, euh, όχι, όχι, ερωτήσεις έχω να κάνω, δεν έχω να κάνω δηλώσεις. Κύριε Επίτροπε, όπως ε, το λέει και το χαρτοφυλάκιό σας, είστε αρμόδιος για, την, ε, για τη φορολογία δεν ξέρω για τα impact assessments όμως. Αυτό το οποίο είπατε εσείς ε, στο Σώμα των Επιτρόπων σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι εσείς έχετε εδώ δύο, με, δύο στα μέτρα και δύο σταθμά. και διαπιστώνω ότι οι προτάσεις που κάνατε εσείς για την ανθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών δεν έχετε προχωρήσει σε καμία μελέτη επιπτώσεων. Και τι χρειάζεται η μελέτη επιπτώσεων για την φορολόγηση των ε, ε, χρηματοπιστωτικών πράξεων όταν εσείς ήδη εκ των προτέρων μας λέτε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι εντελώς άχρηστη μεταξύ τώρα των ε, νέων δημοσιονομικών ε, μέσων, των, των καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων, θεωρείτε εσείς την αλλαγή της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων ως χρηματοπιστωτική καινοτομία. Κυρία Χιούμπνερ, ελπίζω να είναι αρκετά σύντομες οι ερωτήσεις μου και σαφείς για τον Επιτροπό. Καταρχάς ως προς την ε, αντιμετώπιση της φορολόγησης ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα κατά τρόπο που να καλύπτονται και εταιρείε που δεν ανήκουν στον τομέα αυτών ή, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητες χρηματοπιστωτικές στις οποίες δεν εμπλέκεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας καν. Ή θα μπορούσατε ενδεχομένως να σκεφτείτε κάποιες ε, ε, οικονομικές δραστηριότητες να αποκλειστούν από αυτόν τον ε, φόρο. Δεύτερη ερώτηση. Ακούμε συζητήσεις για τα ευρωομόλογα από πολύ σημαντικούς ε, φορείς και προσωπικότητες, ειδικού και λένε ορισμένοι ότι είναι δυνατόν υπό την ισχύουσα συνθήκη, ενώ κάποιοι λένε όχι δεν αρκεί η ισχύουσα συνθήκη, χρειάζεται νέα, χρειάζεται τροποποίηση. Έχει Επιτροπή τουλάχιστον εξετάσει εάν είναι δυνατή, δυνατή εισαγωγή ενός ευρωομολόγου υπό την υφιστάμενη συνθήκη. Κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι δεν απαντήσατε πολύ σωστά την ερώτηση και το ερώτημα των Ελλήνων για το ότι είπατε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Είπατε ότι είναι στο χαρτοφυλάκιο του όλοι Ρεν και όχι στο δικό σας. Ναι, αλλά είσαστε συλλογικό όργανο στην Επιτροπή και μαζί κάνετε τη δουλειά που κάνετε. Και μια και ακούγονται και διάφορες επικρίσεις, εκείνοι οι οποίοι είναι κατά του ευρωομολόγου ε, λέγεται ότι δεν θέλουν να συμπεριφερθούν κατά τρόπο φιλοευρωπαϊκό, να στηρίξουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτό να δούμε και να το σταθμίσουμε μέσα στην όλη συζήτηση. Επίσης, λέτε ότι είσαστε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα. Καταλαβαίνω τη θέση αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την επόμενη κήρυξη τη επιτροπή σε μια πράσινη βίβλο, γιατί όλα αυτά θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να αναπτύξετε non-papers, στα οποία παραδείγματι να λέτε ότι υπάρχουν εναλλακτικέ εναλλακτικέ μία, δύο, τρει να τι καταγράψετε και έτσι να ξεκινήσει μια συζήτηση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει καθόλου τεθεί επιτάπητος είναι η ε, αποξήρανση εντό εισαγωγικών των φορολογικών οάσεων. Το έχουμε εξετάσει αυτό καθόλου. Έχει σκεφτεί κανεί μήπω υπάρχει εκεί κάποια λύση. Είναι δυνατόν ενδεχομένω κάποιε Ελβετίε ή νήσοι κτλ. να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Θέλουμε να το πράξουμε αυτό. Κύριε Επίτροπε, μία πολύ σύντομη και γρήγορη ερώτηση. Αφορά έμεσα το θέμα το οποίο συζητούμε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τι προθέσεις έχετε για το CCTB? Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, προθεσμίες κτλ. Πώς έχει δεσμευθεί η Κομισιόν. Λάρς. Λάρς. Ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο. Οπότε θα κάνω δύο σύντομες δηλώσεις και θα θέσω ένα ερώτημα. Ο διακεκριμένος επίτροπός μας είπε ότι επιζητεί τη μη μετακύληση του φόρου στους καταναλωτές. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω διότι βάσει των μελετών δεν υφίσταται τέτοιος φόρος επί της γης που να μην μετακυλίεται. Ο διάβολος, όπως λέμε στα αγγλικά, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πού ε, κρύβεται ο διάβολος? Στη στρέβλωση. Αν κάνετε υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις, θα έχετε πολυάριθμες στρεβλώσεις και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτό το ευκταίο και ε, ρωτώ το εξής ε, το ενδεχόμενο της επιβολής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συνδέεται μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες οποιοδήποτε εταιρικού ζώου. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ Εάν θέλετε να αποφύγετε ως επιτοπλίστων της τρευλώσης αγοράς, ε, θα πρέπει να επικεντρωθείτε και στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των ε, ε, φορέων που δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μπορείτε να τους σχολιάσετε παρακαλώ. Η Πρόεδρος, θα μπορείτε να κάνετε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σε απάντηση των, στις των συναδέλφων. Δεν έχω πολύ χρόνο. Ας σχολιάσω το CCTV γιατί μου υποβάλλετε διάφορα ερωτήματα. Θα υποβάλλουμε ε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 πρόταση, δηλαδή είναι στα τελικά στάδια προετοιμασίας η πρότασή μας ε, και Λίαν, συντόμως ε, θα έχετε επιτάπητος συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής. Ως προς την αξιολόγηση αντικτύπου, όπως το σχολίασε και η κυρία Περές και άλλοι συναδελφοί της, αληθεύει αυτό που είπατε στον τομέα αυτό και σε προηγούμενες θητείες του Κοινοβουλίου. Γνωρίζω, κυρία περέσο ότι προεδρεύατε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και γνωρίζετε πόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα της φορολόγηση και απαιτεί διεξοδική αξιολόγηση αντικτύπου, διότι συντρέχει ανάγκη αξιολόγηση ταυτόχρονη των διαφόρων φορολογικών βάσεων για να δούμε με ποιο τρόπο οι διάφορες βάσει θα επηρεάσουν ε, τις αγορές, ε, τις πληθυσμιακές ομάδες ε, και ούτω Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να πάρουμε στα τυφλά μία απόφαση. Αυτό κάνουμε λοιπόν, κάνουμε μία ενδελεχή αξιολόγηση αντικτύπου στην Επιτροπή και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουμε αυτό τον αρχικό στόχο. Ε, ο αρχικός πολιτικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι η τελική απόφαση ε, θα ε, πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Όχι, εμείς θα σας υποδείξουμε μέσα από την πρότασή μας ποια είναι η σωστή ρότα, ποια είναι η σωστή οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη γνώμη μας. Ε, σχετικά τώρα με το χρηματοπιστωτικό τομέα και το θέμα των στοιχείων των ενεργητικού και των χρεογράφων, ε, κοιτάξτε, όταν οικοδομούμε συγκεκριμέ... Ε, μάλλον σχεδιάζουμε συγκεκριμένε προτάσει, οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύψουμε και αυτή τη διάσταση της equity για να προβλέψουμε ενδεχόμενες εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις που θα χρειαστούν κατά πάσα πιθανότητα ούτως ώστε να είναι δίκαιοι οι φόροι που επιβάλλουμε. Προφανώς αν διαπιστώσουμε ότι ε, προκύπτει κάποιο πρόβλημα, θα εξετάσουμε προτάσεις για να μετριάσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα οποιοδήποτε μέτρου. Ε, για τους φορολογικούς ε, παραδείσους, η καλή οικονομική, φορολογική συγγνώμη, διακυβέρνηση εν γέννη είναι η απάντηση. Ήδη ε, το Δεκέμβρη θεωρώ ότι σημειώθηκε πρόοδος διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε πολιτική συγκατάθεση για την διοικητική συνεργασία στα φορολογικά θέματα. Τούτο είναι ένα στοιχείο της, ε, του πακέτου χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης ε, και ε, με την Ουγγρική Προεδρία τώρα συζητούμε κάποια άλλα στοιχεία του πακέτου, κάποιες σχετικές οδηγίες, συμφωνίες διμερείς με τρίτες χώρες κτλ. Πιστεύω ότι η Ουγγρική Προεδρία είναι τουλάχιστον όσο φιλόδοξη όσο και η απερχόμενη Βελγική και θα μπορέσει ε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της ε, να σημειώσει αξιόλογη πρόοδο. Ε, τώρα, για το θέμα των ευρωομολόγων, δεν μπορεί κανείς να παγορεύσει τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων, προφανώς σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στην ακρόασή σα ε, θα συνεχίσετε αυτή τη συζήτηση και συγγνώμη προφανώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταγράψει τις θέσεις σα και την έκβαση των ε, συζητήσεων που γίνονται στο Κοινοβούλιο και θα τα λάβετε όντω υπόψη. Κύριε Μπάκρος. Αναφερθήκατε στο θέμα των στρεβλώσεων. Υπάρχει αυτό το, αυτή η παρενέργεια, αν θέλετε, ε, δηλαδή ε, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ε, απλότητα του φόρου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε να φροντίσουμε και τις διάφορες εξαιρέσεις που χρειάζονται. Και για οποιοδήποτε ζήτημα φορολόγηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένα δίλημα πρώτο οποίο βρισκόμαστε αναγκαστικά. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και θα περάσουμε απευθείας στο επόμενο τμήμα της συνεδρίας μα. Περνάμε στο πάνελ δηλαδή των εμπειρογνωμόνων και έχουμε σημειώσει καθυστέρηση δυστυχώς 20 ε, λεπτών. Ελπίζω να κερδίσουμε πίσω το χαμένο χρόνο, ε, όχι από εσά βέβαια. Θα ακούσουμε πρώτα τον Στέφαν Σολμάιστερ για τα ε, φορολογικά εργαλεία, για τον φόρο του άνθρακα από τον Ζακ Λακασέ και από τον κύριο Βίσκο για τα ε, μη φορολογικά εργαλεία. Σε αυτή, με αυτή τη σειρά σας έχω στον κατάλογό μου, οπότε σας ακούμε με αυτή την ε, σειρά. Ναι. Κύριε Σουρμάιστερ, α, συγγνώμη Επίτροπε, επιθυμείτε να πείτε και κάτι άλλο. Ε, ξέρετε, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν θα μπορέσω να παραστώ στην ε, συζήτησή σας. Έχω ανοιγμένες υποχρεώσεις. Ε, ε, πάντως, συνάδελφοί μου από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ φορολογικών υποθέσεων του ΑΞΟΥΝΤ παρευρίσκονται και μπορούν να συζητήσουν με τους εμπειρογνώμονε και μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάντως για τις πολύ καλές ερωτήσεις και πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά, Πρόεδρος. Ε, μάλιστα, έχει άλλα αυτιά, έχει τους συνεργάτες στο Επίτροπο. Σας ακούει παρότι δεν θα είναι εδώ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Βόλς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να περιορίσω την ε, παρέμβασή μου σε δέκα προτάσεις που θα συμπληρώσουν ορισμένα γραφήματα. Οι προτάσεις μου λοιπόν. Υπάρχει μόνο ένα. Υπάρχει υπερβολική ε, δραστηριότητα σε συναλλαγές, σε ρευστό δηλαδή στις σύγχρονες κεφαλαία λόγω της, βρα... Ε, επί... της κρατούσης κερδοσκοπίας σε πρόθεσμο επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι 87 φορές υψηλότερη αυτή, ο όγκος δηλαδή των συνολικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Μέχρι και 90 φορές μεγαλύτερο ήταν τα τελευταία χρόνια. Μια μικρή ύφεση σημειώνεται λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά στη συνέχεια βλέπουμε ε, πέρσι να παρουσιάσει εκρηκτική ανάπτυξη και αύξηση κατά 30% του παγκόσμιου όγκου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, σε σχέση με την περίοδο πριν από τρία χρόνια στο στην επόμενη διαφάνεια, ακόμη και στις ε, ταχύτερες δραστηριότητες συναλλαγών ε, μπορούμε να σημειώσουμε αποσταθεροποίηση και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών των βασικών προϊόντων και των επιτοκίων και των τιμών των μετοχών, διότι οι τιμές, οι βράχοι πρόθεσμες ενισχύονται από τη χρήση των ε, συναλλαγματικών συστημάτων και σορεύονται σε μακροπρόθεσμες τάσεις. Αυτό το βλέπουμε μέχρι το 2008 με μία σόρευση βραχυπρόθεσμη και συνεχή των τάσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που εκφράστηκε και μέσα από τα μηχανογραφημένα συστήματα συναλλαγών και που αποτέλεσε τελικά την μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι ακόμη και σε δεδομένα πέντε λεπτών, βραχυπρόθεσμα δηλαδή, σημειώνω εδώ στην τρίτη μου διαφάνεια, την τάση η οποία χαρακτηρίζει τελικά την, ε, το, το σύστημα αυτό και το οποίο αξιοποιεί τελικά το σύστημα ε, μεγάλη συχνότητα όπως ονομάζεται, High Frequency Trading System. Στην επόμενη διαφάνεια, καλό παράδειγμα θα ήταν το να δούμε την εξέλιξη από 60 σε 150 δολάρια της τιμής του πετρελαίου μέσα σε 18 μόλις μήνες με ένα παράδειγμα το οποίο ε, υπογραμμίζει πως αυτή η ακραία ανάπτυξη τιμής του πετρελαίου χαρακτηρίζεται από την σόρευση βράχη πρόθεσμων ε, αυξήσεων λόγω της ε, μεγάλης κερδοσκοπίας στις τιμές αυτές. Στην επόμενη διαφάνεια οι τιμές των μετοχών επίσης χαρακτηρίζονται από μία αλληλουχία αυτά που ονομάζουν ε, οι συναλλασσόμενοι σχηματαγορές bull market και bear market είτε στις ΗΠΑ είτε στο ΗΠΑ Βασίλειο είτε στη Γερμανία. Επομένως η υπερβολική συχνότητα δεν είναι εξαίρεση αλλά είναι το κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών. Και στην τρίτη μου θέση και διαπίστωση, αυτή η υπερβολική αύξηση των κύριων και πιο σημαντικών τιμών ευνοεί τις δραστηριότητες ε, εισοδηματικού χαρακτήρα περισσότερο, απόδοσης δηλαδή περισσότερο και εμποδίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην πραγματική ε, οικονομία. Δεν αναπτύσσονται δηλαδή επιχειρηματικές δραστηριότητες και έτσι ουσιαστικά αυτή η υπερδραστηριότητα και το υπερβολικό βραχυπρόθεσμο κέρδος παρεμποδίζει την πραγματική οικονομία, ε, οικονομική ανάπτυξη. Αντίστοιχα βλέπουμε μέσα από την περίοδο της υποτίμησης, η οποία οφείλεται στην υπερβολική ανάπτυξη των τιμών των μετοχών, των βασικών αγαθών και της στέγης, αυτή την υπερβολική ανάπτυξη να την ακολουθούν ε, χαράδρες, δηλαδή σημεία σημαντικής πτώσης των αντίστοιχων τιμών αυτών των τριών κατηγοριών προϊόντων. Για να περάσω τώρα στα ομόλογα. Η Ελλάδα πριν από ένα χρόνο είχε, είχε επιτόκιο 6,5%. Μέσα σε τέσσερις μήνες μόλις, μόνο με την ενίσχυση του πριμ του CDS, έφτασε σε 12%, σε 12% επιτόκιο για τα ομόλογα. Έτσι ώστε να φτάσει τελικά το Μάιο του 2010 στο Ταμείο Διάσωσης όπως ονομάστηκε και στην επόμενη ε, διαφάνεια βλέπουμε την ε, ίδια μοίρα για τα Ιρλανδικά ομόλογα και ξέρουμε ότι θα τα ακολουθήσουν και τα Ισπανικά και τα Πορτογαλικά. Γιατί. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Είναι τόσο κερδοφόρο που η Deutsche Bank ή η Allman ή όποια, όποιος άλλος οργανισμός δεν πρόκειται να το αφήσουν ανεκμετάλλευτο. Είναι αυτοί οι κανόνες του παιχνιδιού που τους επιτρέπουν την υπερβολική κερδοφορία. Και έτσι φτάνω στην πρόταση παριθμών 5. Ένα μικρό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 0,05%. Οι πέντε μονάδες βάσης δεν θα επηρεάσει όλες τις συναλλαγές που στόχο θα έχουν την διαφύλαξη, την διατήρηση δηλαδή, των ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων του ενεργητικού. Το ίδιο ισχύει και για το hedging, για την αντιστάθμιση, γιατί και ο αντισταθμιστής διαφυλάσσει τις θέσεις του. Εάν δούμε παραδείγμα τη μετοχή σε τιμή 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει κανείς τη συναλλαγή 2,5 ευρώ μόλις. Τώρα μόλις δύο λεπτά μου έχουν, θα, θα ζητήσω ακόμα. Λοιπόν, ένας ε, φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα ενισχύσει σημαντικά το κόστος εκείνων των συναλλαγών που δεν έχουν αντίκτυπο, που δεν έχουν μάλλον αντιστοιχεία στην αγορά. Όσο πιο υψηλή είναι η κερδοφορία, τόσο πιο υψηλό και το κόστος που θα επιβάλλει αυτός ο φόρος. Και έτσι φτάνω και στο 7 στι προτάσεις μου, ότι ένας τέτοιο φόρο θα, σημάνει σημαντική, θα επιβάλλει σημαντική ε, εισφορά από εκείνου του παράγοντε, των οποίων οι δραστηριοτήτε έχουν σημαντικά συμβάλει στην ανάπτυξη αυτή τη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση το 2008-2009. Και ταυτόχρονα αυτοί οι χρηματοπιστωτικοί παράγοντε, οι οποίοι ακόμη επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση πραγματική οικονομία, αυτό που μερικέ φορέ ονομάζεται boring banking, βαρετή ε, δραστηριότητα, τραπεζική δραστηριότητα, δεν θα επιβαρυνθούν. Γιατί ε, βέβαια αυτός ο φόρος δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ των ε, τραπεζών, ε, μάλλον ένα γενικό φόρο για τι τράπεζε δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των τραπεζών οι οποίε ενισχύουν την πραγματική οικονομία και εκείνε οι οποίε ασχολούνται μόνο με την κερδοσκοπία. Ενώ ο FTT, ο φόρο δηλαδή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα μπορεί να στοχεύει ειδικά τι τις ε, κερδοσκοπικέ αυτέ δραστηριότητε. Έτσι φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημαντικό έσοδο περί τα 30% ε, με βάση τα δεδομένα του 2007 στην, στην πρόταση υπαριθμών 9 ε, δεν αποτελεί σημαντικό τεχνικό πρόβλημα εισαγωγή ενό τέτοιου φόρου και υπαριθμών 10 ότι μπορεί ένα τέτοιο φόρος να αποτελέσει τον κύριο υπερεθνικό ευρωπαϊκό φόρο και τελικά τον πρώτο παγκόσμιο φόρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο Ζακ Λεκασέ τώρα για το φόρο για τις εκπομπές άνθρακα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω από την εξή διαπίστωση. Πρόκειται για μια δουλειά που εδώ και λίγο καιρό, την, ε, εδώ και σχετικά μάλλον αρκετό καιρό την ε, κάνουμε. Για το θέμα για τη φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακος δεν είναι ακόμα τόσο καθαρό. Ε, το βασικό πιο είναι ότι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν επαρκούν και θα ήθελα να κάνω ορισμένες απλές προτάσεις. Πρώτη διαπίστωση, η φορολόγηση της ενέργειας στην Ευρώπη δεν αυξήθηκε, μειώθηκε από τις αρχές του 2000, πράγμα το οποίο είναι αντιφατικό με τους ε, στόχους που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Δεύτερον, η αγορά του διοξιδίου σίγουρα μας επιτρέπει να ορίσουμε μία τιμή εκπομπών για τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν καλύπτει παρά μόνο το 40% των ρηπαντικών εκπομπών και η τιμή που έχουμε στην αγορά είναι πάρα πολύ ε, χαμηλή και ασταθείς για να μπορέσει να μας οδηγήσει σε μία ε, δραστηριότητα σταθερή. και οι τιμές ε, δεν είναι οι σωστές κυρίως όσον αφορά στον τελικό καταναλωτή. Θα σας πω μερικά για τον τελικό καταναλωτή αργότερα. Η πρόταση θέλει να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα και αυτό προς δύο κατευθύνσεις. Η αγορά του ε, άνθρακα υφίσταται, δεν μπορούμε εμείς ε, να την εμποδίσουμε να λειτουργήσει ικανοποιητικότερα και αυτό αυξάνοντας ε, την ε, τιμή, μειώνοντας δηλαδή τις ποσότητες των ποσοστώσεων που διοχετεύουμε στην αγορά. Δεύτερον, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας που ανέφερε ο Επίτροπος, αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε Η αύξηση όμως των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος προέρχεται κυρίως από τις μεταφορές και επίσης μεγαλύτερο μερίδιο το έχουν οι οδικές μεταφορές, εμπορικές ή αστικές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τιμή της παροχής ενέργειας δεν είναι επαρκώς υψηλή σήμερα για να παίξει καταστατικό ρόλο και για το θέμα των διατάξεων για τις εκπομπές των αυτοκινήτων είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν μας επιτρέπει αυτό να λύσουμε το πρόβλημα η παραγωγή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων στα αυτοκίνητα, όχι τις εκπομπές. Άρα καταναλώνεται λιγότερη βενζίνη και το κόστος μεταφοράς μειώνεται. Και αυτό δεν παίζει κατασταλτικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να θεσμοθετήσουμε στα σύνορα ένα τέλος ε, διοξιδίου του άνθρακος για να μπορέσουμε να στείλουμε στον τελικό χρήστη ένα μήνυμα, ένα μήνυμα σαφές. Και επίσης ε, για το θέμα ε, των, ε, της φορολόγησης των εκπομπών, τα εισαγόμενα προϊόντα δεν υφίστανται σε αυτό το φόρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και να το λύσουμε, διότι υπάρχει, υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων που παράγονται εντός της, εσωτερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Εσωτερικής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η εισφορά στα σύνορα πιστεύω, αυτό το τέλος στα σύνορα πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα μπορούσαμε θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε δύο τρόπους, είτε το τέλος στα σύνορα, είτε τη φορολόγηση των εισαγωμένων προϊόντων, το οποίο, πράγματα τα οποία είναι απόλυτα συμβατά με τους κανόνες της ΠΟΕ. Ο Επίτροπος είπε προηγουμένως δε ότι θα πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τα φορολογικά συστήματα, ούτω ώστε να στοχεύει η φορολόγηση στην κατάσταση τα πολέμηση των κακών συμπεριφορών και την ενθάρρυση των καλών συμπεριφορών. Αυτά είναι πράγματα που ισχύουν για τη φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήταν όμως ιδιαίτερα κρίμα η Κομισιόν να μην μελετήσει γενικώς την γενική φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακος. Ο Επίτροπος είπε ότι πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα πολύπλοκο και με μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις. Είναι επικίνδυνο να διατυπώνουμε εμείς κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σήμερα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κρατούν λογιστική για το, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα ενισχυθεί αυτή η τάση στο μέλλον. Θα πρέπει, αν θέλουμε να έχουμε κάτι το, κάτι το θετικό ε, στο μέλλον ε, για το, θα πρέπει να έχουμε φορολόγηση εισαγωγών, εξαγωγών αλλά και τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να υπόκειται και αυτός επιπτώσεις του φόρου. Ευχαριστώ, κύριος Βίσκο, Βινσέντο Βίσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ για να κερδίσω χρόνο θα σας διαβάσω ένα σύντομο σημείωμα στα Ιταλικά. Έστειλα όμως ε, στα Αγγλικά στην Επιτροπή ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να το διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται. Η ύφεση και η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 οδήγησαν σε μία αύξηση των ελλημάτων, των δημοσίων ελλημάτων σε όλα τα κράτη και αυτό λόγω των αυτομάτων επιπτώσεων, σε επιπτώσεις των εσόδων των κρατών μελών και λόγω των πράξεων υποστήριξης και σωτηρίας των τραπεζών. Στην Ευρώπη η κρίση των εθνικών προπολογισμών διακύβευσε την ίδια την δημοσιονομική σταθερότητα και το ενιαίο νόμισμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει ότι στις προθυμένες οικονομίες για το 2011 θα αυξηθεί το δημόσιο χρέος κατά μέσο όρο κατά 29 πόντους του ΑΕΠ με πιο γάλλες διακυμάνσεις στο 40% και το 2014 ή ο σταθμισμένος μέσος όρος θα ξεπερνάει το 100% σε αυτές τις ε, χώρες. Πάντοτε το, Διεθνέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι αν ο στόχος των οικονομικών πολιτικών θα ήταν να φτάσει το δημόσιο χρέος το 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2030 θα χρειαζόταν να έχουμε μία διόρθωση των προϋπολογισμών κατά 8 9 μονάδες του ΑΕΠ. Θα έπρεπε επίσης να προσθεθεί και μία επιπλέον διόρθωση 4-5 ε, πόντων σε ορισμένες χώρες για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των συντάξεων και των ε, εξόδων υγείας. Για τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα πολύπλοκο trade-off μεταξύ εξυγίανσης των δημοσιονομικών και οικονομικής ανάπτυξης. Η εξυγίανση θα απαιτούσε περικοπές ή μπλοκάρισμα της οικονομίας και σε ορισμένες περιπτώσεις και αποπληθωρισμό. Αυτό όμως θα καταδίκαζε τις χώρες μας σε μια παρατεταμένη στασιμότητα και σε υψηλή ανεργία για πάρα πολλά χρόνια που δεν θα άφηναν ε, κατά μέρο καμία χώρα. Η Γερμανία ας πούμε. Το 60% των εξαγωγών της Γερμανίας γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις οικονομίες δηλαδή οι οποίες θα επλήττονταν από αυτά τα μέτρα και θα, θα οδηγούσαν σε ύφεση λοιπόν και την γερμανική οικονομία. Και σχετικά με το Hellcat. Θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστιες επιπτώσεις σε όλο το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα. Στις χώρες μας λέγεται ότι θα πρέπει να μειωθεί το έλλειμμα των, ε, του δημοσίου χρέους, σαν να ήταν το χρέος υπεύθυνο το οποίο δημιούργησε την κρίση. Και άμα συνεχίσουμε ακόμη παραπάνω από αυτήν την, την κρίση θα αυξηθεί και το χρέος. Πιστεύω ότι η κρίση θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί μέσα από συλλογικές δράσεις. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να απολευθερώσουμε τους δημόσιους προϋπολογισμούς από το έξτρα χρέος το οποίο συσσωρεύθηκε λόγω της κρίσης και να τους ε, να τους ξαναφέρουμε στην λογιστική κατάσταση του 2007 και θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο στο οποίο τα κράτη θα μεταφέρουν την ποσόστοση του κυρίαρχου χρέους που δημιουργήθηκε το 2007 μετά από την κρίση. Και εκεί αναγνωρίζεται η ίδια υπόσταση των συλλογικών χρεών. Και θα δίνεται και σχετική εγγύηση. Επίσης, θα πρέπει να γίνει φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών πράξεων, οι οποίες να... και η φορολόγηση αυτή να χρησιμεύει για την απόσβεση του χρέους προς το συγκεκριμένο ταμείο. Στη συνέχεια, τα ποσά τα οποία επιστρέφονται στο ταμείο θα πρέπει να μετατρέπονται σε ενεργά κεφάλαια. Επίσης, το Ταμείο θα πρέπει να κεφαλαιοποιεί τις ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας 3 και αυτό θα οδηγούσε στην δημιουργία κερδών. Και αυτό θα βοηθούσε στην εξισορρόπηση των χρεών και θα έδινε ελευθερία στα δημοσιονομικά των κρατών μελών και θα απέφευγε και τον κίνδυνο ενός γενικού αποπληθωρισμού. Το ρίσκο θα τον αναλάμβανε ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος όμως θα κέρδιζε και από την παρουσία στην αγορά ενός νέου χρήστη, ο οποίος θα ήταν ιδιαίτερα ισχυρός κυρίως από τα έσοδα που θα ε, συσσόρευε από αυτή τη νέα φορολόγηση. Ας πούμε στην Νότιο Κορέα υπάρχει ένας ειδικό φόρος για τις εισαγωγές στη χώρα που χρησιμεύει για την κεφαλοποίηση των τραπεζών. Εγώ αυτή την πρόταση την ξεκίνησα πριν από έξι μήνες μαζί με τον καθηγητή Πλά και τον, κύριο, τον καθηγητή Ντασέγκελ βασιζόμενος και στις θέσεις του Μάριου Μόντι για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, αλλά και βασισμένος στο σχέδιο των κυρίων Γιούνκερ και Τρεμόντι. Η πρότασή μου αφορά αυτό το έξτρα χρέος που δημιουργείται από την κρίση και που είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Εμένα η πρότασή μου δημιουργεί τα περιθώρια για αυτόνομη φορολογική πολιτική. Και τα ευρωμόλογα πιστεύω ότι θα βοηθούσαν να χρηματοδοτηθεί το χρέος. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις τράπεζες να κεφαλαιοποιηθούν και αυτές που δεν θα το καταφέρουν θα πρέπει να πτωχεύσουν. Οι προτάσεις μου λοιπόν είναι πολιτικές. Να βρεθεί μια συνεργατική απόφαση μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το οποίο όμως εμάς μας φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Η Άννη Ποδηματά και ο Ούντο ναι, θέλουν να μιλήσουν. Η Ντανίτα, κάποιος άλλος παρακαλώ. Άννη τότε. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομη γιατί πραγματικά είμαστε απελπιστική κατάσταση. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ Σάρον. Λέει η κυρία Ποδήματα, ε, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Κύριε Σουλμάιστερ, πολύ ε, ε, αξιόλογα και αξιοπερίεργα αυτά τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε κυρίως για τις ε, εξελίξεις τα τελευταία χρόνια του χρηματοπιστωτικού τομέα σχετικά με το είδος δηλαδή των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών που οδήγησαν σε αυτήν την ε, διόγκωση άνευ προηγουμένου των του όγκου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τέλος πάντων, περνάω στην ερώτησή μου απευθείας. Με ποιο τρόπο κατά τη γνώμη σας μπορούμε να εισαγάγουμε ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγοντας ε, τον ε, κίνδυνο της επανακατανομής ε, που, στον οποίο αναφερθήκατε. Κύριε Κασέ, εν συντομία θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η ιδέα για την εισαγωγή ενός μεθοριακού συνοριακού φόρου άνθρακα πρέπει να εγκριθεί πρώτα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Έτσι δεν είναι. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση αυτού του είδους ο φόρος θα μπορούσε να θεσπιστεί χωρίς πρωτήτερα να προβούμε σε κάποιο είδους εναρμόνιση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δηλαδή πρώτα να έχουμε εισάγει ένα είδος φόρου άνθρακα ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Βίσκο, για τα ευρωομόλογα και πάλι εδώ ε, θα ήθελα να σχολιάσω την αντεπιχειρηματολογία που υπάρχει. Πώς ανταπαντάτε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι τα ευρωομόλογα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδεχομένω μεγαλύτερο κίνδυνο και να διαβιβάσουν πλημελές μήνυμα κυρίως προς τις χώρες που ε, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αυτή την εποχή. Πώς απαντάτε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι ο κίνδυνος με τα ευρωομόλογα είναι η αύξηση των επιτοκίων ενάρετων προϊόντων. Γιατί χρησιμοποιούμε θρησκευτικού όρους τώρα τελευταία. Ε, τα ευρωομόλογα ε, μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη αύξηση των επιτοκίων και μείωση των επιτοκίων για τους αμαρτωλούς, για τα αμαρτωλά προϊόντα σε σχέση με τα ενάρετα. Πρόεδρος. Θα ακούσουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε πια χρόνο. Ούντο, Ντανούτα και Φιλίπ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλου του εμπειρογνώμονε για τη συμβολή του στη συζήτηση. Μα έχουν βοηθήσει πολύ να προχωρήσουμε στην συζήτηση. Και θα ήθελα για να συμπληρώσω τα όσα είπε και η συγγήτριά μα, για τον κύριο Σουλμάιστα, για, τους διάφορους, ε, για τα διάφορα φορολογικά μέσα που βρίσκονται υπό συζήτηση. Θα ήθελα να μου πείτε εάν βλέπετε διαφορετικές τάσεις ή ε, πτυχές καθοδήγησης θα έλεγα των διαφόρων αυτών φόρων. Γιατί δεν έχουμε μόνο την, ε, τα έσοδα αλλά και την πίεση που μπορεί να ασκήσει ένας φόρος σε μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, ε, το πώς μπορεί να καθοδηγήσει δηλαδή, την αγορά. Σε αυτό μπορείτε να μας κάνετε κάποια σχόλια, Ντανούτα Χούμπνερς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ στον κύριο Σουλμάιστερ να απευθύνω μια ερώτηση και να συζητήσουμε λίγο περισσότερο το συσχετισμό μεταξύ του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και της κερδοσκοπίας. Στην πέμπτη σας πρόταση αναφέρετε, αναφέρεστε στον κίνδυνο και τα χρηματοπιστωτικά παράλογα, ε, παράγωγα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παράγωγα μπορούν να εκφραστούν και σε όρους υποστήριξης που προσφέρονται για τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες. Δηλαδή μπορούν να προστατεύσουν τις τράπεζες από τον αυξανόμενο για το μέλλον ενδεχομένω κίνδυνο. Γιατί λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί τα παράγωγα τα κρίνεται μόνο ως κερδοσκοπικά μέσα, ως μέσα κερδοσκοπίας. Και δεύτερη ερώτηση με το φορό χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μας λέτε ότι θα έχουμε υψηλότερο κόστος συναλλαγών, αλλά μέσω συμπληρώνεται λέγοντα ότι το υψηλότερο κόστος ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει επερχόμενες κρίσεις. Ξέρουμε όμω από την εμπειρία μας, ε, από τέτοια, ε, από τις κρίσεις αυτές, ότι δεν εξασφαλίζεται ε, προστασία από τις φούσκες τις χρηματοπιστωτικές. Πού στηρίζετε λοιπόν αυτή η διαπίστωση. Φίλιπ, ε, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις που με απασχολούν και εμένα και που ακούστηκαν από άλλους ε, συναδέλφους. Απλώς για τον κύριο Σουλμάινστερ για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών FTT. Ακούστηκε ότι αν το εισαγάγει αυτό ω μέτρο η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη τη και την ακολουθήσει ο υπόλοιπο κόσμο, θα είναι σαν να αυτοπυροβολείται, ε, δηλαδή θα επιβαρύνει μόνο τη δική τη οικονομία και όχι του άλλου. Από την άλλη κάποιοι λένε ότι αυτό πρέπει να εισαχθεί μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Εάν δεν είναι εφικτή δηλαδή η επιλογή του φόρου αυτού ω ε, εφαρμόσιμου σε ολόκληρη την Ευρώπη των 27 κρατών μελών, μπορεί να επιβληθεί μόνο για την ε, ζώνη του ευρώ. Δεύτερη ερώτηση, και πρέπει να πω ότι με εκπλήσει αυτό που διαβάζω μέσα στο εγγραφό σας, ότι προτείνεται όχι ευρωομόλογα, αλλά παγκόσμια ομόλογα. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα, αλλά εάν αναγνωρίσετε κι εσείς ο ίδιος ότι δεν είναι η πιθανότερη εξέλιξη προς την οποία πηγαίνουμε για τα επόμενα, τους επόμενους μήνες ή χρόνια ενδεχομένως, και αν μας μιλάτε στην πρόταση σας για τις προτάσεις Τρεμόντι και Γιούνκερ και τις ε, μπλε ή κόκκινες μετοχές, ή μάλλον τα μπλε ή κόκκινα ομόλογα. Ε, ξέρουμε ότι αυτή η τάση τώρα τα παγκόσμια ομόλογα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Ή μάλλον δεν θα υλοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Αν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί δεν θα είναι στο εγγύς μέλλον. Ε, τότε τι έχετε να μας προτείνετε εναλλακτικά για τα μπλε ή τα κόκκινα ομόλογα και τις προτάσεις Γιούνκερ και Τρεμόντι που είναι επιτάπητος, που είναι προς συζήτηση, γιατί εγώ βρίσκω ότι είναι πολύ πιο εφικτές, έστω και αν χρειαστεί πολλή προσπάθεια και μεγάλο ε, άλμα πίστης θα έλεγα από όσους πρόκειται να τα εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και θα αποτολμήσω και εγώ μια δική μου ερώτηση για τον κύριο Σουλμάιστα. Στο πρώτο μέρος της ε, παρουσίας σας ουσιαστικά απαντάτε στα επιχειρήματα ορισμένων οικονομολόγων ότι μπορεί να ε, επιταχυνθεί η δραστηριότητα των συναλλαγών ή να ενισχυθεί η ρευστότητα στις αγορές και ότι αυτό είναι καλό πράγμα από την εξαγωγή του φόρου. Εν πάση περιπτώσει όμως από την παρουσία σας, εγώ θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Εάν έχουμε ταχύτερες συναλλαγές, οι κύκλοι αλλαγής θα πρέπει και οτι αυτο ειναι καλο πραγμα απο τους του φορου εν παση περιπτωσει ομως απο την παρουσια σας εγω θα ηθελα να επισημανω το εξη εαν εχουμε ταχυτερες συναλλαγες οι κυκλοι αλλαγης θα πρεπει και αυτη να ειναι πιο σύντομοι. Έτσι δεν είναι. Εσείς μας λέτε όμως ότι ίσως είναι πιο μακροπρόθεσμη αυτή η κύκλη εξέλιξη. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες εξηγήσεις, αλλά μάλλον γραπτό τα έλεγα, μήπως προσπαθήσετε να το αναλύσετε εδώ. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτή η, η κυκλική τάση όταν έχουμε ε, συναλλαγές υψηλής συχνότητας, και μια κάποια, ένα κάποιο εύρος χρονικό σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους, ιστορικές περιόδους, μήπως τελικά δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μόνο μια αλλαγή συχνότητας σε μια συνολική διακύμανση. Η οποία τελευταία ανάλυση θα ήταν αναμενόμενη δεδομένως της συχνότητας των συναλλαγών. Και τώρα για να περάσουμε στα απαντήσεις θα παρακαλέσω να δοθούν οι απαντήσεις με τη σειρά που ακούστηκαν από τους ε, συναδέλφους μας. Κύριε Σουλμάιστερ. Σας ευχαριστώ για το, την πρώτη ερώτηση. Ποιες συναλλαγές ενδεχομένως οδήγησαν ε, σε, αυτό, σε αυτή την ε, ανευπροηγουμένου ε, αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Βάσει της Τράπεζας των Διεθνών Διακανονισμών, 58% των συναλλαγών τα τελευταία τρία χρόνια οδήγησαν σε αυτή την αύξηση και ε, πρόκειται φυσικά για συναλλαγές υψηλής συχνότητας, ε, κυρίως στην αγορά συναλλάγματος. Οι συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος οδήγησαν σε αυτή την αύξηση. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για αυτό το φαινόμενο και βασιζόμαστε σε στατιστικούς αλγορίθμους που αποπειρούνται να ε, διερευνήσουν κάποιες ε, βραχυπρόθεσμες παρατυπίες. Τι σημαίνει ιδιαίτερα ε, βραχυπρόθεσμες παρατυπίες, κάποια δευτερόλεπτα σημαίνει. Δεν υπάρχουν πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. 20 hedge funds τις είπα παραδείγματος χάρη μόνο. Ε, και πρόκειται για κάτι που γίνεται στους βασικούς σερβες. Ε, δηλαδή, αν είσαστε κοντά στο σερβερ, στη βασική ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου, έχετε ένα χιλιοστό το δευτερολέπτο περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλους συναλλασσόμενους και αυτό είναι καταπληκτικό πλεονέκτημα. Και όσο αυξάνεται η ταχύτητα ε, των συναλλαγών, τόσο λιγότερο μπορούμε να λάβουμε υπόψη θεμελιώδεις παραμέτρους ε, τη αγορά και δυσχεραίνουν τα πράγματα. Οι οικονομολόγοι, οι ακαδημαϊκοί δεν χρησιμοποιούν αυτέ τι έρευνε. Σε κυρίως ε, εγώ παρατηρώ τη συμπεριφορά τους και τι διαπιστώνω ότι ε, όσοι έχουν αυτές τις πληροφορίες έχουν μόνο ένα δευτερόλεπτο για να τις χρησιμοποιήσουν και ήταν πολύ χαμηλότερο το έλλειμμα στη ΣΥΠΑ σε σχέση με το αναμενόμενο. Έχουν κλάσματα δευτερολέπτου για να αντιδράσουν μόνο και ποτέ δεν μπορούν να δημιουργήσουν ποσοτικοποιημένες προσδοκίες για τις συναλλαγές. Δεν μπορούν να πούν ότι βάσει των πληροφοριών που έχουμε θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά είναι ανοησίες, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες, αλλά... Ε, έχουμε λοιπόν το θέμα των ευλόγων προσδοκιών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την θεωρία για να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο. Δεύτερον, είπατε είναι δυνατή εισαγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν υιοθετηθεί αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σχετικά απλό το σύστημα. Γιατί, διότι το ζήτημα, ε, θέμα συμψηφισμού και διακανονισμών ε, λειτουργεί ηλεκτρονικά ε, και ακόμη και για τις έξω χρηματιστηριακές συναλλαγές ε, μελλοντικά θα πρέπει να περάσουμε από μια κεντρική πλατφόρμα αντισυμβαλωμένων, έτσι ονομάζεται. Βέβαια θα, δυσκολέψει το πράγμα αν έχουμε ε, πολλαπλές ε, πλατφόρμες. Αλλά ε, ε, πώς θα γίνει η μετανάστευση όλων των συναλλαγών σε μία πλατφόρμα. Κοιτάξτε, βασικό στοιχείο είναι 24ωρη βάση των συναλλαγών και η μετανάστευση, του immigration, αφορά σε συναλλαγές που γίνονται στην ίδια... στην ίδια χρονική ζώνη ε, και το, θα πρέπει βέβαια να διαπιστώσουμε αν θα μπορέσει να υπάρξει επαρκής ανταγωνισμός με την εισαγωγή ενός τέτοιου ε, φόρου. Τέλος, Όλα είναι συνάρτηση της συνολικής αξιολόγησης του οικονομικού αντικτύπου όλων αυτών των εξαιρετικά βραχυπρόθεσμων ε, συναλλαγών. Α, το κατά πόσο συνδέονται με βασικά μεγέθη οικονομικά, βάσει της εμπειρίας μας, ε, εξαρτάται από τις αποκλίσεις που σημειώνονται από την βασική ισορροπία. Δηλαδή, βάσει της θεωρίας περί ισορροπίας, εάν μία αγορά δεν μπορεί να σπρώξει την τιμή ενό ε, στοιχείου του ενεργητικού προς την κατεύθυνση ε, της ισορροπίας ε, για να υπάρχει ισοδυναμία πόλη, της τιμής πόλης αγοράς και αντίθετα εκτοξεύεται ανωδικά ή καθοδικά, τότε τι έχουμε αγορές ανωδικές ή καθοδικές, η bull market και η bear market αλλά αυτό διαφέρει πολύ από τον κόσμο των οικονομικών μεγεθών γενικότερα. Αν θεωρείτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών ε, οπωσδήποτε θα αποσταθεροποιήσουν την αγορά γιατί δεν χρησιμοποιούν βασικά οικονομικά μεγέθη, δηλαδή πληροφορίες για την προσφορά και για τη ζήτηση, τότε τι σημαίνει αυτό ότι 25% των συναλλαγών θα θα μετατοπιστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίσως αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό και θα καλό θα ήταν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το καθήκον, να στο θέσω έτσι, του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή την εξυπηρέτηση τη ε, πραγματική οικονομία. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι σημαντικέ οι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Ο κύριο Μπούλμαν μας ε, ρώτησε για τα εφορολογικά κίνητρα εδώ υπάρχουν τέσσερα διακρίσεις ανάμεσα σε ένα τραπεζικό τέλος και ένα τέλος επί συναλλαγών. Ένας τραπεζικός, ένα τραπεζικό τέλος συνδέεται με ένα συγκεκριμένο απόθεμα. Γι' αυτό το λόγο ε, και κάπου τοποθετείται μέσα στον ισολογισμό της τράπεζας. Άρα εξορισμού, εκφύσεως δεν μπορεί να τιμωρήσει ε, τις ε, συναλλαγές. Πρέπει να συνδέει το φόρος με μια οικονομική ροή. Αυτή είναι η βασική συναλλαγή ανάμεσα στο φόρο επί των συναλλαγών και το φόρο επί κάποιων θέσεων του ισολογισμού τραπεζικών και άλλων ιδρυμάτων. Για τα παράγωγα τώρα, προφανώς δεν είναι κάτι κακό εκφύσεως τα παράγωγα. Τα παράγωγα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο. Μια αεροπορική εταιρεία, παραδείγματο χάρη, αναμένει ότι ε, θα αυξηθεί ενδεχομένω η κυροζήνη. Οπότε ε, αγοράστε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο και αν σημειωθεί όντω αυτή η αύξηση του καυσίμου, τότε αντισταθμίστε εσεί τον κίνδυνο, διότι έχει αναβαθμιστεί και η αξία του προθεσμιακού σα συμβολέου. Αλλά η αξία των συναλλαγών επί είναι τέτοια ώστε να μην μπορούμε να εισαγάγουμε ε, ε, κανένα μέτρο ποσοτικό. Δηλαδή, ε, μην ξεχνάτε τι γίνεται στο γερμανικό χρηματιστήριο. Συγγνώμη, ναι, το ξέρω ότι βιάζεται, αλλά τι να κάνω για μου λέτε να απαντήσω. Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε τις υπόλοιπες απαντήσεις σε γραπτός, γιατί είναι και πολύ τεχνικά αυτά τα ζητήματα και δεν έχουμε και χρόνο. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συζήτηση, αλλά έχετε τη δυνατότητα να στείλετε γραπτός τις απαντήσεις σας. Εντάξει. Uh, uh, Επιτρέψτε μου να απαντήσω και εγώ με τη σειρά μου στις ε, ερωτήσεις που αφορούν ε, την φορολογία του άνθρακα. Από τις δύο ερωτήσεις θα ξεκινήσω από τη δεύτερη. Είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο τύπου εναρμόνιση, πιστεύω, ε, της φορολογίας για τον άνθρακα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μέρος του συλλογισμού. Διότι ένα από τα διδάγματα των τελευταίων ετών είναι ότι εάν στηριζόμαστε στις επιλογές των επιμέρους κρατών, στην εισαγωγή δηλαδή στα επιμέρους κράτη, της φορολογίας των άνθρακα και η Γαλλία δεν αποτελεί καθόλου καλό παράδειγμα τότε και λόγω της εσωτερικής φορολογικής ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προχωρήσουμε καθόλου. Άρα χρειάζεται κάποιου τύπου ευρωπαϊκή φορολογία ή κάποια μορφή εναρμόνιση της φορολογία των εκπομπών του άνθρακα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να δώσουμε και το σωστό μήνυμα και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό. Όπως είπα και νωρίτερα. Δεύτερο, θα ήταν αυτό συμβατό με τους κανόνε του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εδώ πιστεύω ότι εάν ε, διαβάσετε προσεκτικά το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή τις δηλώσεις του Πασκαλαμή πέρυσι για τους ειδικού φόρους ε, για τον άνθρακα, η απάντηση είναι ναι, είναι συμβατή εφόσον εισαχθούν κατά τρόπο σωστό, δηλαδή χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων, ε, υπό την έννοια αυτών που καταγράφονται μέσα στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Άρα και πάλι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στρέβλωση τιμών ως προς την συμπερίληψη άνθρακα σε διάφορα προϊόντα και δεν αρκεί η φορολόγηση της ενέργειας. Ναι, αποτελεί απαραίτητο, ε, απαραίτητο αναγκαίο δηλαδή βήμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φορολόγηση της ενέργειας, πλην όμως δεν είναι επαρκές, διότι υπάρχει η παρέκκληση του εμπορίου, δηλαδή η σημαντική αύξηση της εισαγωγής προϊόντων με σημαντικά ποσοστά άνθρακα, σημαντική επιβάρυνση άνθρακα. Λοιπόν, αν αυτό προστεθεί στο σύνολο των ευρωπαϊκών εκπομπών, συνολικά δεν μειώνονται οι ε, εκπομπές, η επιβάρυνση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μάλλον μένει σταθερή και τελικά δεν επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος αυτής της ειδικής φορολογίας. Εγώ θα απαντήσω ε, μαζί στις δύο απαντήσεις. Πρώτη και τελευταία. Την πρώτη και την τελευταία. Τι προτείνω για τις διάφορες προτάσεις που έχουν τώρα υποβληθεί. Μα οποιαδήποτε πρόταση σαν αυτή του Γιούνκερ Τρεμόντι που επιτρέπουν να βάλουμε στον κοινό κορβανά το ευρωπαϊκό χρέος πρέπει να υποστηριχθούν. Τώρα, η δική μου πρόταση θεωρεί ότι η πρόταση Juncker Τρεμόντι είναι συμπληρωματική. Στόχος είναι να απολευθερώσουμε τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, την φορολογική πολιτική των κρατών μελών, από το άχθος των διορθώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στην πλάτη του λαού. Φτιάχνουμε λοιπόν εμείς αυτό το κοινό καλάθι όπου ενώνουμε το χρέος και συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως πριν. Σταματάμε όμως τις σπατάλες επανερχόμενοι δηλαδή στη δημοσιονομική κατάσταση του 2007 η πρόταση Γιούγκερ Τρεμόντι μόνη της μπορεί να είναι προβληματική. Αν βρεθούν με αυτό το χρέος και τα blue bonds και τα red bonds, ε, για τα κόκκινα ομόλογα μπορούν να επιβαρυνθούν σημαντικά. Οπότε θα ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες Πιο συγκεκριμένα οι γαλλικές, οι γερμανικές, οι βελγικές, οι ολλανδικές και οι άγγλικες ε, κατέχουν μεταξύ του 15 και του 20% του ΑΕΠ τους ομόλογα των πιο αδυνάμων χωρών. Αν η πρόταση Γιούγκερ Τρεμόντι κολλήσει με αυτούς τους τίτλους, τότε θα μπλοκάρει όλο το χρηματο... ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι θα πρέπει να αγοράσουν στην τιμή της αγοράς. Στη δική μου την περίπτωση ε, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, διότι αυτά τα παίρνουμε, τα μετακινούμε, τα βάζουμε αλλού και αυτό χρηματοδοτούνται. Εγώ 30 χρόνια τη ζωή μου έχω κάνει πολιτική. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μην βρίσκει κανείς συμφωνία. Αλλά πρέπει να έχουμε συνέστηση γι' αυτό. Εμείς για τα επόμενα 5-6 χρόνια βρισκόμαστε σε απόλυτη στασιμότητα και επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τον πολίτη. Και μετά από αυτά τα 5-6 χρόνια θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συλλογικά και συνεργατικά, γιατί από αυτό έχουμε να κερδίσουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τόντι πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη διέξοδο από την ε, τωρινή από τα τωρινά προβλήματα και να μην ε, προξενούμε νέα Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά πολλά θέματα για συζήτηση σήμερα. Ε, και θα παρακαλέσω, αν έχετε γραπτά σχόλια, ε, να μας τα διαβιβάσετε πιο αναλυτικά σχόλια ενδεχομένως, Σας σα περιμένουμε, θα περιμένουμε με αδημονία. Και περνώ στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το υπαριθμό 4. Μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των διεθνών επενδύσεων. με τον κύριο David Κάσα, εισηγητή. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση για το μέλλον των, ε, της πολιτικής των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα ασχολείται με τις διμερείς συνθήκες, με τις διμερείς επενδύσεις. BITS ονομάζονται, bilateral δηλαδή investment treaties, και δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα των ξένων, άμεσων ξένων επενδύσεων, άξε. Έχουν γίνει κάποιε συζητήσει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή την αποκλειστική αρμοδιότητα μπορεί να την ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πιο σαφής η κατάσταση όταν συζητήσουμε αναλυτικές προτάσεις οι οποίες ε, θα στηρίζονται σε ε, ιδέες για ρύθμιση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διμερών αυτών διεθνών ε, συμφωνιών διμερών αυτών συμφωνιών επενδύσεων. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με εσωτερικές και με εξωτερικές επενδύσεις οι οποίες έχουν υποφελείς ε, επιφελή αντίκτυπο για την απασχόληση μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξωτερικές επενδύσεις μπορεί να έχουν άμεσα αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένους τομείς ή περιοχές, αλλά οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι δεδομένο ότι έχουν ε, να προσφέρουν μόνο ωφέλη και θα ήταν σκόπιμο να προσελκύουμε στο δυνατόν περισσότερες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι δε Ευρωπαίοι επιχειρηματίε θα πρέπει να, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει να επενδύουν στο εξωτερικό μόνο όταν είναι βέβαιο ότι η επένδυσή του είναι ασφαλή και προστατευμένη, δηλαδή μέσα σε ένα σταθερό, υγιέ και προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον. Οι συμφωνίε που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν ήδη, θα πρέπει βεβαίω να τηρηθούν και θα πρέπει να τεθεί επαρκή χρόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε αυτή να διατυπώσει τι νέε συμφωνίε που θα αντικαταστήσουν σταδιακά όλες τις διμερείς συμφωνίε συμφωνίες για επενδύσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ισχύσει ε, μία ενιαία και ομοιόμορφη λύση για τους πάντες και θα πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε ε, συμφωνίας, τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων παραγόντων και την εξέλιξη στην ανάπτυξη των οικονομικών μας εταίρων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διαφυλαχθεί και η έννοια της ασφάλειας, της προβλεψιμότητας και να αποφευθεί ο υπερβολικός γραφειοκρατικός φόρτος, να μην επιβληθούν δηλαδή υπερβολικές ε, υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη. Σε κάθε στάδιο θα πρέπει αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι συμφωνίες και οι διαδικασίες να είναι ε, εφικτές και οι, ισχύ, οι τωρινές διαπραγματεύσεις, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις να μην ανατραπούν. Επικεντρώνομαι λοιπόν στα πιο σημαντικά θέματα, στις προτάσεις μου. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει μια γενική συζήτηση για το μέλλον, για τις μελλοντικές επενδύσεις και ότι θα μπορέσουμε τελικά να Ε, δώσουμε λύσεις για τις επενδύσεις. Εγώ θα κάνω τις προτροπολογίες μου όταν θα έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι όλοι θα συνεργαστούμε μαζί για να συζητήσουμε το θέμα αυτό κατά τρόπο σοβαρό και επικοδομητικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Jean-Luc Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ως και εισηγητής ε, των σοσιαλιστών θα πάρω το λόγο. Ευχαριστώ για αυτήν την ε, παρουσίαση τον εισηγητή. Εμείς έχουμε μία διπλή και σημαντική πρόκληση για να βελτιώσουμε την απασχόληση και να προωθήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων χωρών. Εμείς έχουμε πάρα πολλές τρέχουσες συμφωνίες. 3.000 συμφωνίες από το 1959 και μετά και είχαν ως στόχο την ε, διασφάλιση, ως στόχο τη διασφάλιση των μη διακρίσεων προ και μετά των επενδύσεων, την προστασία των επενδυτών, το, την, δικαστική, την νομική προστασία των επενδυτών τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε και νομικά να έχουν την νομικά και νομοθετικά να έχουν την διασφάλιση οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Εμείς θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια διεθνή συμφωνία επενδύσεων, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μοιρασμένη αρμοδιότητα μεταξύ κομισιών και κρατών μέλων. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δε ότι μετά από τη Λισαβόνα οι άμεσες εξωτερικές επενδύσεις εντάσσονται στην εμπορική πολιτική που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να κρατήσουμε ε, να, να, να κρατήσουμε ενωμένε τις, πράξεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Θα πρέπει εμείς να προστατεύσουμε τις επενδύσεις ε, που θα γίνονται στις τρίτες χώρες. Δεν θα πρέπει ο κόσμος πλέον να χωρίζεται μεταξύ αναπτυσσομένων, αναπτυγμένων χωρών και αναπτυσσομένων χωρών. Θα πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη να κρατάει προστατευτικές ε, θέσεις θα πρέπει να ευνοεί επίσης τις αηφόρες επενδύσεις σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο και αυτό ανάλογα με τις, σύμφωνα μάλλον με τις οδηγίες της όξε. Επίσης είναι θεμελιώδης η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, σύμβαση για την επίλυση διαφορών με τους πολίτες τρίτων χωρών, διότι δεν συμμετέχουμε εμείς ακόμα σε αυτήν τη σύμβαση. Πρέπει να ορίσουμε λοιπόν εμείς την ευθύνη αμφωτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να τοποθετηθώ για αυτό το σχέδιο για να δώσω και κάποιε ιδέε στον κύριο Κάζα. Ε, και ε, για τη μελλοντική συνεργασία με τους συνεισηγητές. Από τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας και βάσει του άρθρου 286 η πολιτική άμεσων ξένων επενδύσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, με θετικό τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και προστατεύονται καλύτερα μέσω προτύπων οι επενδύσεις. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Συμφωνώ με τις προτάσεις του εισηγητή και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποιες άλλες. Στην πρώτη παράγραφο για την έλλειψη προβλεψιμότητα τη συνθήκη θα ήθελα να παρατηρήσω το εξή. Στη συνθήκη Λισαβόνα δεν υφίσταται ορισμό σχετικά με το τι είναι ακριβώ οι ε, ξένε άμεσε επενδύσει. Επίση, ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πρότυπα προστασία για να μην υπάρχουν ε, παραθύρακια για ερμηνεία του νόμου από ε, τα δικαστήρια διαιτησίας, ε, γιατί σήμερα διακρίνονται από χαρακτηριστική έλλειψη διαφάνειας. Επίσης, οι εθνικές διμερείς συμφωνίες επενδύσεων θα ήθελα να προσθέσω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσως όρου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, και αυτό θα είναι εφικτό γιατί θα καλύπτω από τον ίδιο ΦΠΑ και από τα ίδια πρότυπα. Είναι ένα νέο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τέλος, ε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τις Ευρωπαϊκές Επενδυτικές Συμφωνίες αναμένεται μικρότερος κίνδυνος, μεγαλύτερη ε, ασφάλεια όπερ και θα ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να κάνουν ε, επενδύσεις στην αλλοδαπή. Φυσικά πρέπει να εισακουστούν κατά τη διάρκεια των δεπραγματεύσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άρα υποβάλλω και κάποιες σχετικές τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Υπάρχει άλλος κοιόδης που θέλει να παρέμβει. Α, ο Πασκάλ. Oui, merci. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να παρέμβω και ένα-δύο θέματα πολύ στόμα για την εκθέση αυτή. Σημαντικό, μα φαίνεται, εφόσον υπάρχει συζήτηση να εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα τη αμοιβαιότητα, θα θέλαμε στην έκθεση αυτή να εισαχθεί η έννοια τη αμοιβαιότητα. Είναι θέμα επικαιρότητα, έχει πολιτικό αντίκτυπο σημαντικό και στηρίζουμε αυτή την πρόσφατη δράση τη Επιτροπή. Δεύτερο στοιχείο, οι συμφωνίες επενδύσεων ενσωματών το σύνολο των ε, πολιτικών της ε- Ένωσης και όχι μόνο τις εμπορικές αλλά και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτικές και ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως υπόθηκε νωρίτερα, καλό θα ήταν ενδεχομένω να επανεπεξεργαστούμε τους μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν πλέον όλους αυτούς τους πολιτικούς στόχους ε, στην, ε, στο συλλογισμό πάνω στον οποίο στηρίζονται. Αυτά είχα να πω εγώ ως ιδέες για τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριε Κάτσα, θέλετε να επανέλθετε σε τίποτα συγκεκριμένο. Ναι, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν. Πρόκειται για έκθεση ιδέα πρωτοβουλία, όπως πρέπει να υπενθυμίσω. Μόνο 1500 λέξει επιτρέπονται και άρα μπορούμε βεβαίω να συμπεριλάβουμε τις προτάσει που ακούστηκαν σήμερα, αλλά θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο από την ομάδα των φιλελευθέρων που είπε ότι ο επακριβής προσδιορισμός της ξένης επένδυσης, ελοδοπή επένδυση, δεν προβλέπεται και γι' αυτό χρειάστηκε εγώ να το συμπεριλάβω θα χρειαστεί να το συμπεριλάβω στην έκθεση που θα ακολουθήσει. Και άρα θα δώσουμε στη συνέχεια αυτόν τον ορισμό. Πάντως καλό είναι να διευκρινίσουμε αυτούς τους όρους. Τα σχόλια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον να βρίσκουν σύμφωνο. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει όμως να περιμένουμε την ε, γνωμοδότηση για το θέμα αυτό που είναι πιο συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Προθεσμία για τις τροπολογίες 17 Ιανουαρίου, συζήτηση 7 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 28 Φεβρουαρίου και στην κατουσία αρμόδια, καθήλυνα αρμόδια των Ιανουάριο για να πάει στην Ολομέλεια τον Μάρτιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προς το παρόν για την ε, έκθεση αυτή. Είπε και ο Ντέιβιτ ότι έχει κανένα δύο ακόμη γνωμοδοτήσεις και άρα θα έχουμε να ξανασυστήσουμε μαζί του το σημείο 5 για τις ρυθμίσεις, για τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να μονοπολώ το χρόνο ομιλίας. Ήθελα να σας πω απλώς ότι δύναμη της ε, συνθήκης Λισαβόνας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ε, συνιστούν πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό φυσικά στα πλαίσια της κοινή εμπορικής πολιτικής. Έχοντας τούτο κατά νου, καλωσορίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποσκοπεί στο να ε, χειριστεί το προσωρινό στάδιο των εξελίξεων. Δηλαδή, ε, έχουμε τώρα κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι τρίτε χώρες αφενός και συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι τρίτε χώρε αφετέρου. Ε, και το σχέδιο γνωμοδότησής μου αποπειρά να διευκρινίσει τις ε, αναφορές που γίνονται άμεσε ξένες επενδύσεις ε, σε ολόκληρη τη συνθήκη, οδηγώντας σε ένα συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας των άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 Ιουλίου 2010. FDI είναι το ακρονίμιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις ε, στα αγγλικά και το οποίο χρησιμοποιεί στην στη γνωμοδότησή μου. Για μείωση του γραφειοκρατικού άκθους, μειώνοντας τον την περίοδο αναμονής, ε, που θεωρείται ε, υπερβολική. Επίσης, σε βασικό στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου οι επενδυτές θα έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις επενδύσεις τους. Έχουν συμπεριλάβει ρήτρες, χάρη στις οποίες η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ε, κάποια σαφή στοιχεία αν μα δώσει τη διευκρινήση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφαιρέσω αυτά τα στοιχεία από το σχέδιο γνωμοδότηση. Επίση, ε, προσπαθώ να διευκρινίσω σε ποιε περιπτώσει μπορεί να ανακαλέσει την άδεια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει μια χώρα, μια διμερή συμφωνία για τι ε, ε, διμερείς επενδύσεις. Επίσης άλλο θέμα είναι μορφότυποι που μπορούν να χρησιμοποιούν και ο θελός στα κράτη-μέλη προς διευκόλυνση ε, αυτών των διμερών ε, επενδυτικών συναλλαγών των BITS. Ε, επίσης, προσδιορισμός των βελτίστων ε, πρακτικών ε, βάσει των υφιστάμενων συμφώνων επενδύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύσκολα θα μπορέσει να ανακαλέσει τις ισχύουσες συμφωνίες ε, για να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκές συμφωνίες. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται και τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε ε, να διαπραγματευτεί ενδελεχώς ε, την έκβαση τέτοιων επενδυτικών διαπραγματεύσεων που θα είναι προς όφελος και των κρατών μελών και των επενδυτών. Ε, προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία που με τους σκιώδεις συγητές ελπίζω να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για αυτό το θέμα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όπως γνωρίζετε. Πρόεδρος, μάλιστα. Εγκαίρος πρόλαβα να σηκωθώ για να, ξανα... για να ανοίξω το μικρόφωνο και να προεδρεύσω. Ε, κάποιος άλλος σκιώδης. Α, ο Thank you very Ευχαριστώ ε, κάποιες ιδέες, δύο-τρεις ιδέες ε, θα σας ε, εκθέσω για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις με τον εισηγητή. Λοιπόν, ο στόχος είναι να έχουμε προσωρινές ε, ρήτρες σχετικά με τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, ε, ενώ δεν υπάρχει ακόμη κοινή τέτοια πολιτική. Ε, στο μεταξύ θα διατηρηθούν ενισχύ αυτές οι συμφωνίες ή μπορούν να συναυθούν και άλλες νέες, αν λάβουν την άδεια, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ποιο ο σκοπός ε, αυτού του εγχειρήματο. Ε, οι συμφωνίες δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν πρέπει να επικαλύπτονται από ευρωπαϊκές συμφωνίες και ούτε και να συνιστούν φράγμο κατά την, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μελλοντικών εμπορικών πολιτικών τη Ένωση. Γι' αυτό το τελευταίο στοιχείο ο κ. Κάζα προτείνει κάτι και θα ήθελα τώρα ακριβώ να συζητήσουμε αυτή τη ε, διαγραφή που έχει κάνει ο κύριο Κάζα, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώ για ποιο λόγο το έκανε. Επίση, ε, πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα προσωρινά μέτρα, για λόγο, θα, ε, για πόσο, πόσο χρόνο θα διαρκέσουν. Στο έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνεται αρχική περίοδο ισχύω πενταετή και η Επιτροπή ΙΝΤΕ αντιπροτείνει τέσσερα χρόνια. Και εγώ πιστεύω ότι τα πέντε χρόνια είναι υπερβολικά μεγάλη περίοδο, αλλά ο εισηγητή δεν υπέβαλε καμία τροπολογία επ' αυτού ήθελα λοιπόν να συζητήσω μαζί του για αυτό το θέμα, ούτω ώστε να ε, καταλήξουμε στο ευλογότερο χρονικό διάστημα. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία με του ε, λοιπούς και τους εισηγητές και τον εισηγητή μα, τον κύριο Κάζα, ούτω ώστε να ε, φορήσουν οι προσπάθειές μας ε, στον τομέα των επενδύσεων. Ε, Πασκάλ και μετά ε, ο Ούντο. Δεν βλέπω να παίρνετε το λόγο, άρα ο Ούντο παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο σκιώδης ηγητής είναι ο κύριος Μπέρμαν εκ μέρους ομάδας μου, δεν μπορούσε όμως να έρθει σήμερα εδώ για να συγχαρεί τον κύριο Κάσα, να δώσει τα σχόλιά του. Υπάρχουν κάποιες πτυχές πολύ σημαντικές εδώ. Καλωσορίζω λοιπόν τις προτάσεις του κύριου Κάζα και θα ήθελα να φροντίσουμε όταν υπάρχουν νέες αρμοδιότητες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε και στη θέση να ορίζουμε, να δίνουμε ένα νέο κοινό ορισμό να είμαστε στη θέση να προτείνουμε ένα νέο κοινό ορισμό του τι εννοούμε ως ξένες άμεσες, άμεσες ξένες επενδύσεις. Άξε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πάντοτε η επιχειρηματολογία μα στηρίζεται στο ότι οι αλλαγέ που θα γίνουν σε αυτέ τι διμερεί συμφωνίε θα πρέπει να στηρίζονται στη λογική μια ε, ορθολογική εξέλιξη, προστασία του περιβάλλοντο, κοινωνικών προδιαγραφών. Και αυτές θα είναι και κάποιες από τις προτάσεις που θα καταθέσει ο σκιώδης συγκητής μας. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Κάποιο άλλο παρακαλώ. David, θες να, να eh, Δεν θα μιλήσω πολλή ώρα. Έχω ήδη στον μιλήσει με τον σοσιαλιστή συνάδελφο. Συμφωνώ με τις προτάσεις του, όπως άλλωστε συμφωνώ και με τις προτάσεις του συναδέλφου των φιλελευθέρων για την τροπολογία υπαριθμών Εδώ προτείνω τη διαγραφή του κειμένου. Και αυτό γιατί είναι πολύ ασαφές το κείμενο όπως είναι διατυπωμένο. Θα ήθελα να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο για τον επενδυτή όταν γίνεται λόγος λοιπόν για την πρόταση αυτή και διαβεβαιώ τους συναδέλφους πώς θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό και αυτή την παράγραφο δηλαδή έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν χρειάζεται να το απαλείψω από την πρότασή μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τις δύο αυτές προτάσεις με τον χρόνο έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και πάλι 17 Ιανουαρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, συζήτηση 7 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 28 Φεβρουαρίου και στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή το Μάρτιο, όπως άλλωστε και στην Ολομέλεια θα πάει το θέμα στο Μάρτιο, τουλάχιστον έτσι λέει το χρονοδιάγραμμα προς το παρόν και προχωρώ τώρα στο σημείο υπαριθμών 7-6 της ημερήσης διάταξης, εταιρική διακυβέρνηση χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης από, την Ashley Fox, από τον Ashley Fox. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα να τον πιο σύντομο και θα ξεκινήσω ευχαριστώντα του λοιπού συγκητέ, του σκιώδη συγκητέ δηλαδή, οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτήν την ε, πρόταση. Βέβαια, δεν είχα επαρκή ε, περιθώρια χώρου και έτσι δεν μπορούσα να συμπεριλάβω όλε τι προτάσει. Πάντω, ευχαριστώ και την κυρία Προσέσκη και την υπηρεσία τη για την υποστήριξη που μα έχουν προσφέρει στην υπόθεση αυτή. Δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ, αλλά πάντω την ευχαριστώ. Έχω συζητήσει πολλέ φορέ ε, με του συναδέλφου, με χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με εποπτικέ αρχέ, με την Επιτροπή. Και μετά από όλε αυτέ τι συζητήσει καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η κύρια προσέγγιση, η βασική μου προσέγγιση θα είναι η αρχή της προσαρμογής ή της επεξήγηση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία ε, τέτοια προσέγγιση και αν κοιτάξουμε από τις ΗΠΑ τη σχετική εμπειρία, η αυστηρά ρυθμιστική τους προσέγγιση δεν τους προστάτευσε από την τελευταία κρίση. Περισσότερο από ότι κάποια άλλη προσέγγιση και γι' αυτό πιστεύω ότι μόνο ει βάρο των χρηματοπιστωτικών μας οργανισμών θα ήταν το να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε του Αμερικανού σε αυτή την προσέγγιση. Πιστεύω κράταντα πω ο, ο είναι ενσωματωμένος αλλά και απαραίτητο για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Το πρόβλημα μπορεί, τα προβλήματα μάλλον μπορεί να προκύπτουν όταν κανείς άκρατα προ, αναλαμβάνει κινδύνους και ανεξέλεγκτα. Και γι' αυτό κάποιες από τις προτάσεις μου στόχο έχουν να δράσουν διορθωτικά ως προς τη συμπεριφορά αυτή. Επίσης, μπορούμε να έχουμε μια κατάλληλη στρατηγική για, την, ε, για τον προσδιορισμό του κινδύνου και για τον έλεγχο από πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, ακόρες της όρεξης του οργανισμού αυτού. Η ε, εταιρική διακυβέρνηση λοιπόν μπορεί να είναι ικανοποιητική εφόσον είναι κατάλληλα και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν να την εφαρμόσουν. Χρειάζεται ναι. λοιπόν να έχουμε σε κάθε χρηματοπιστωτικό οργανισμό υπεύθυνα άτομα με ναι ικανότητες, με πείρα, με ηθική ακαιρεότητα. Δηλαδή το τρίγωνο της πείρας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και του ακέραιου χαρακτήρα. Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς κίνδυνο στην επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και να μην, μην ανησυχούμε. Ως προς αμοιβές. Έχουμε ένα παράδειγμα του CRD3, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε, γιατί ήταν λάθος. Και ω προ τι εποπτικέ αρχέ, ελληνικούς μηχανισμού κλπ. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρωταρχικό του ρόλο είναι η ακρίβεια, η εξέταση δηλαδή για αξιολόγηση, αν είναι ακριβή τα στοιχεία που δίνονται. Δεν πρέπει λοιπόν αυτόν τον αυτόν τον ρόλο να τον επιβαρύνουμε με επιπλέον καθήκοντα που έχουν να κάνουν με κρίσει αξιολογικέ. Πιστεύω ότι χρειάζεται πεστρός διάλογος, αλλά θα πρέπει να είναι τριμερής. Εποπτικές αρχές, ελεγκτικές αρχές και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να συμμετάχουν σε αυτόν. Ο δε μέτοχος και ιδιαίτερα ο θεσμικός μέτοχος θα πρέπει να λαμβάνει και αυτός ενεργό ρόλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον προσδιορισμό στρατηγική του και στην λογοδοσία για τη στρατηγική αυτή και ενισχύει έτσι την συμμετοχή σε μια γενική συνέλευση των μετόχων που πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτική διότι θα ήταν βέβαια και άσκοπη αλλά και ανέφικτη. Γι' αυτό πρόεδρε σταματώ. Θεωρώ ότι οι κοινέ τροπολογίε με άλλους συναδέλφους ε, θα ήταν χρήσιμε ε, στους τομείς που είναι δυνατόν να υποπληθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Άσλεϊ Φόξ για τη δουλειά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους κοιόδης εισηγητές κατά την εκπόνηση του σχεδίου γνωμοδότησης έλαβε υπόψη πολλές καλές ιδέες παραδείγματο χάρη σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας, το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και ούτω καθεξής. Ε, μπορούμε να διευκρινίσουμε την περαιτέρω κάποια επιμέρους στοιχεία της έκθεσης. Και το σημαντικό είναι να έχουμε μία ομοιόμορφη προσέγγιση σχετικά ε, με τον corporate tax, τον εταιρικό φόρο. Δεν είναι θετικέ οι εξελίξει δεδομένες τη χρηματοπιστωτικής καταιγίδα που βιώσαμε. Ε, κάποιες ε, τέτοιες συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων και άρα δεν ε, θα ισχύσουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Θα ήθελα λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύψουμε κάποια ημιτελή στοιχεία και θα συζητήσουμε τον εισηγητή για αυτά τα στοιχεία. Οι επόπτες παραδείγματος χάρη πρέπει να ενισχύσουμε την, το ρόλο τους για τη διαχείριση του κινδύνου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των συμφωνιών περί της διαχείρισης και αντιστάθμισης αναβάθμισης των κινδύνων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχουν στη διάθεσή τους ε, οι επόπτες ε, όσοι ευθύνονται για τη διαχείριση των κινδύνων πρέπει να έχουν ενισχυμένο ρόλο τόσο ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και αμερόληπτα. Ε, κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οπωσδήποτε ο ρόλος του να αξιολογηθεί από κάποιο εξωτερικό φορέα διότι έχει ευρύτατες αρμοδιότητες ε, ε, κάθε διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιολογεί τον κίνδυνο κάθε διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, για την αποζημίωση ως προς τους κινδύνους, ε, αυτό το κομμάτι της έκθεσης θα πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε με άλλες εκθέσεις που έχουμε ήδη εγκρίνει στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται επικάλυψη ούτε επαναλήψεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι μέρος ενός συνολικού πακέτου. Κατόπιν, χρειάζονται διευκρινήσει σε σχέση με τι προσδοκίε μα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια πράσινη βίβλο και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενδέχεται να αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε. Ποιε είναι αυτέ και πώ ιεραρχούνται οι προτεραιότητέ μα. Θα υποβάλω εγώ τροπολογίε για κάποια από αυτά τα στοιχεία που ανέφερα, αλλά για μια σειρά ερωτημάτων πάντω θεωρώ ότι δεν θα δυσκολευτούμε να καταλήξουμε σε συμφωνή και με επικοδομητικό τρόπο θα καταλήξουμε σε μια ε, καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ έχει ζητήσει τον λόγο. Καλημέρα. Δεν μπόρεσα να συμμετέχω στις συνεδριάσεις που μόλις οργανώσατε. Ε, να σας εξηγήσω μερικά για τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Πρώτον, ε, η γενική θέση για την αυτορύθμιση ούτως ώστε να έχουμε κανόνες δημοσίου δικαίου. Ένας από, ένα από τα διδάγματα της κρίσης είναι ότι η αυτορύθμιση δεν ε, λειτουργεί. Πρέπει να έχουμε κανόνες όταν μία τράπεζα ε, παίρνει πολλά ρίσκα ε, και κερδίζει πολλά χρήματα, οι ανταγωνιστές της ε, δεν μπορούν να την ακολουθήσουν ε, και αναμβάνουν άλλου είδου ρίσκα για να κερδίσουν τα αντίστοιχα και είναι τελικά οι πολίτες που την πληρώνουν. <coughs> Αυτό είναι ένα από τα διδάγματα της κρίσης. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Αλχαντράουι ότι θα πρέπει να δούμε με την Κομισιόν τι συγκεκριμένο θέλει να πράξει σχετικά. Δεύτερο, το ρίσκο. Εσείς είπατε ότι η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η διαχείριση του κινδύνου. Πρέπει όμως εμείς να κατανοήσουμε αυτό το ρίσκο και αυτό το ρίσκο δεν εξαρτάται μόνο από την ευθύνη των ενδιαφερομένων αλλά και από τον επόπτη και τους νομοθέτες διότι ένα από τα διδάγματα της ε, κρίσης ε, σε αυτό την πράσινη βίβλο είναι ότι τα ιδιαίτερα πολύπλοκα προϊόντα δεν είναι εποπτεύσιμα και δεν έχει την απαραίτητη κατανόηση ο επόπτης για να μπορέσει να, κατανο... να αξιολογήσει την πραγματικότητα του κινδύνου. Αυτό είναι επίσης ένα από τα διδάγματα της ε, κρίσης, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε. Για την Επιτροπή Κινδύνου ε, χρειάζονται μέτρα και θα υπάρξουν φαντάζομαι κοινέ τροπολογίες για να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των διαφόρων επιτροπών εποπτείας και τις ικανότητες ε, των μελών τους ε, ε, για να μπορούν να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τελευταίο για, τον, για τους κινδύνους θα πρέπει να ενσωματώσουμε και να εντάξουμε και έξω χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, για παράδειγμα, οι κίνδυνοι που είναι δεμένοι με τις κλιματικές αλλαγές. Χρηματοδοτούν οι τράπεζες υποδομές μεταφορών, οι υποδομές ενέργειας κλπ. Θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην απόφαση της, της επένδυσης και το κλιματικό ε, ρίσκο να πραγματοποιούνται ας πούμε Ε, περιβαλλοντικά ε, τεστ ε, stress test για τις υποδομές, αν δηλαδή η υπόθεση ότι θα αυξηθεί η θερμοκρατία, η θερμοκρασία συγγνώμη, κατά 2 ή 3 βαθμούς, τι επιπτώσεις θα έχει κάτι τέτοιο στα θερμοελεκτρικά εργοστάσια ή στους αυτοκινητοδρόμους κλπ. Ε, οι ασφαλιστές είναι οι πρώτοι που πλήγονται από τις αλλαγές ε, του κλίματος ε, και είναι οι πρώτοι που έχουν κατανοήσει ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν προχωρήσει σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να εξετάζεται και αυτό το ρίσκο. Τώρα στην τροπολογία 5, το να βρίσκονται οι τράπεζες μέσα σε ένα board θα πρέπει ή τα διοικητικά στελέχη να έχουν πραγματικές αρμοδιότητες. Θα, διότι στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών δεν υπάρχει ένας ε, ένα πραγματικό αντίβαρο από τη διοικητική πτέρυγα της τράπεζας. Θα πρέπει στις ε, τροπολογίες να περάσει η θέση της Οικονομικής Επιτροπής όπως έτσι είχε ψηφιστεί κατά την συζήτηση του ε, του ΣΕΡ3 πριν τη συζήτηση του Συμβουλίου. Να επανέλθουμε δηλαδή σε αυτήν την αρχική θέση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Μπασέσκου η οποία έχει προβλήματα πτήσεων. και ζητά να τη συγχωρήσετε για την απουσία σας. Η συνεργασία μας ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για την δουλειά του και να πω μερικά πράγματα για τις τροπολογίες μας. Εγώ θα ήθελα, διαβάζοντας το τωρινό σχέδιο, ότι διαβάζω αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν, τα οποία ήδη υφίστανται σε ορισμένες χώρες, σε μία εκ των οποίων γνωρίζω καλά τουλάχιστον. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει απλώς να διαπιστώσουμε ποια είναι η κατάσταση, πρέπει να δούμε πώς να τη βελτιώσουμε. Θα ήθελα να γίνεται μεγαλύτερη αναφορά στο, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας γιατί μιλάμε εδώ συνέχεια για τις εθνικές αρχές. Σίγουρα οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των κανόνων. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους γενικούς κανόνες και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας. Για τα υπόλοιπα προτείνω να ενισχύσουμε λίγο τον έλεγχο, διότι πολλές διατυπώσεις είναι διατυπώσεις καλών προθέσεων που τελικά καταλήγουν στην αυτορύθμιση. Και όπως είπε και ο Πασκάλ, σύμφωνο ως προς τις αρχές τις οποίες διακήρυξε. Um, thank um, Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι η σκιώδης των φιλελευθέρων. Υποθέτω ότι η σειρά μου είναι. Ε, Άσλι, ζητώ συγγνώμη που ε, ε, έκρινες ότι δύσκολα μπορούσες να με παρακολουθήσεις και ότι πότε ήμουν εδώ, πότε δεν ήμουν. Είχα προβλήματα και το ήξερες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για το πλαίσιο που μας δώσατε. Προφανώς μπορούμε να ευσέλθουμε σε λεπτομέρειες, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Μάλλον χρειάζεται κάποια επιμέρους στοιχεία να τα αναπτύξουμε περαιτέρω. Επίσης ε, προκρίνω και εγώ την προσέγγιση της αναλογικότητας. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τι ισχύει για να μπορέσουν να συμμορφωθούν όλοι. Για ε, τα, τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς χρειαζόμαστε αυστηρότερη εφαρμογή και όχι μόνο αυτή η αρχή του and explain. πρέπει να υπάρχουν οι σωστοί μηχανισμοί ελέγχου. Ε, δεν θα ήθελα βέβαια να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό που αναφέρετε στην έκθεσή σας. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί, γιατί ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ε, ότι κανένας δεν θα ασχολείται με την ποιότητα, θα περιορίζεται μόνο στους κανόνες. Κανείς δεν θα ασχολείται με την ευρύτερη εικόνα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Ε, Ούτω ώστε να έχουμε την ευρύτερη εικόνα και να δούμε πώς ε, ε, συνδέονται τα επιμέρους ζητήματα μεταξύ τους και κυρίως να δούμε πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Έτσι, ε, σίγουρα χρειαζόμαστε ποικιλία στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι για πολιτικούς λόγους, δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχουν κάποιοι τις σωστές εμπειρίες, τα σωστά βιώματα, αλλά ε, σε έναν τομέα που τους σπρώχνει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν μας ενδιαφέρουν πολιτικοί προσανατολισμοί, μας ενδιαφέρει το να έχουμε την ευρύτερη εικόνα επίσης. Ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τη, κάποια ε, φρασιολογία που χρησιμοποιήσαμε στην τρίτη οδηγία για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει, ούτω ώστε οι αρμόδιοι να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να λαμβάνουν τις αποφάσεις. Για την πράσινη βίβλο τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται εξής, το εξή ερώτημα. Πρέπει να έχουν αυξημένες ευθύνε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ θα σας απαντούσα καλύτερα να πληρούν τα καθήκοντα που ήδη έχουν και μετά βλέπουμε και έτσι επανέρχομαι σε αυτή την αρχή του κοπλά and explain. Συμμορφώνουμε και εξηγώ γιατί ε, υπάρχουν κάποιοι, κάποια μέλη του Διοικητικού ε, Συμβουλίου που ακολουθούσαν αυτό το, αυτή την έννοια του and explain και δεν τα κατάφεραν. Οπότε πρέπει να δούμε πώς με ευέλικτο τρόπο θα ενισχύσουμε το ρόλο τους ως προς ε, τα, τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που ανήκουν ε, στο μακροοικονομικό σύστημα της χώρας. Ε, είναι πάρα πολύ απασχολημένοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα και άρα ε, αναρωτιέμαι εγώ σε πόσα διοικητικά συμβούλια μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός στα τρία διοικητικά συμβούλια αυτό είναι προσυζήτηση. Δεν θα ήθελα να είμαστε άκαμπτοι και να θέσουμε ένα όριο, αλλά ας απαντήσουμε στο ερώτημα. Θέλετε αυτοί οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν από αριστερά δεξιά και από το ένα συμβούλιο στο άλλο να λειτουργούν ε, ποιοτικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχουμε ποικιλία και να μειώσουμε τα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, καλύτερα κάποιο να έχει ισχυρότατο αξίωμα σε ένα μόνο ε, διοικητικό συμβούλιο, να είναι πρόεδρο σε ένα μόνο συμβούλιο, παραδείγματο χάρη. Για του επιθεωρητέ και του επόπτε, ε, δεν θα έπρεπε να επιβάλλουμε κανόνε και να παρέμβουμε στα λοιπά καθήκοντα των εποπτών ε, ή να καταργήσουμε σχέσει εμπιστοσύνη που ήδη υπάρχουν. Και ξέρετε, στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα μοντέλα διαχείριση και οφείλουμε να τα εξετάσουμε. Και μου έρχεται κατά νου αυτό το ερώτημα. Οι επόπτε δεν πρέπει να ξέρουν ότι κάποιες ε, επενδυτικέ ε, τράπεζες ε, έχουν τεράστια ποσά σε κάποιους κρεμείς υπεράκτιους λογαριασμούς, παραδείγματος χάρη. Δεν πρέπει αυτό να τεθεί υπόψη των εποπτών τέτοιου είδους πράγματα ε, χρειάζονται απάντηση και οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πώς συνδέονται αυτά τα επιμέρους ζητήματα μεταξύ τους. Επίσης, ε, για τις ψηφοφορίες ε, υπάρχουν οι κανόνες για αποκάλυψη των πληροφοριών, κυρίως για τους θεσμικούς επενδυτές. Εγώ έχω το δικό μου κατάλογο με τα πράγματα που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και αυτό είναι ένα από αυτά. Ε, σχετικά με το πακέτο εποπτικής αρχιτεκτονικής που βλέπουμε στη ρήτρα αναθεώρησης ε, και ε, βάση των πρακτικών σύγκλησης των αρμοδίων αρχών, προβλέπεται αξιολόγηση μεταξύ άλλων της σύγκλησης ως προς την λειτουργική αυτονομία των εποπτικών αρχών και των προτύπων που αντιστοιχούν στα πρότυπα της εταιρική διακυβέρνησης. Αντιστοιχεί λοιπόν ανάμεσα στις αρχές και στις εταιρικέ αρχές. Νομίζω και αυτό το θέμα θα πρέπει να το πραγματευτούμε μέσα στην έκθεση, δηλαδή οι βέλτιστες πρακτικές ε, που αναμένουμε στον τομέα της εταιρική διακυβέρνησης ε, μέσα στους θεσμικούς ε, φορείς, νομίζω αναγκαία μα οδηγούν σε μεταρρυθμίσει ε, στην γενικότερη αρχιτεκτονική και του συστήματο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, και καλό θα ήταν να δούμε τι προβλέπεται ήδη στι ρήτρε αναθεώρηση για του θεσμικού επενδυτέ. Και μην ξεχνάτε την συνάντηση που έχουμε προγραμματίσει ε, για αυτή την εβδομάδα. Αυτά δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να παρέμβει. Όχι, ο Άσλι λοιπόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που έλαβαν όλη τη συζήτηση. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι προσπαθείτε να, πει, να χρόνο, άλλα σχόλια δεν θα κάνω παρά μόνο ότι θα ξανασυζητήσουμε και όταν έχουμε τις ε, τροπολογίες στα χέρια μας θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ λέει, κυρία Μπόιλ. Πραγματικά πολύ σύντομη επέμβαση. Τώρα θα πρέπει να δω αν θα μπορούσα να ανακαλύψω κάπου τον ε, Υπουργό στου διαδρόμου. Σε πάση περιπτώσει όμω έχουμε 17 Φεβρουαρίου, 28, 16 Μαρτίου φορεί και στην Ολομέλεια, τον Απρίλιο στην πρώτη σύνοδο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και προχωρούμε τώρα για να ακούσουμε τον απερχόμενο εκπρόσωπο ή τον απελφέντα καλύτερα εκπρόσωπο της Προεδρίας τον κύριο Ρέντερς. Μείνετε στη θέση σας, παρακαλώ. Okay, 10 ε, λεπτά διάλειμμα θα έχουμε μέχρι να φτάσει ο υπουργό Ρίντερ, γιατί ξέρετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με την βελική πολιτική. Σε δέκα λεπτά ε, θα επανέλθουμε. questions. Right, well, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, που περιμένατε τόση ώρα και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά όλοι οι πολιτικοί είμαστε και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα θέματα και στον προπολογισμό ιδιαίτερως. Με χαρά λοιπόν τώρα καλωσορίζω για άλλη μια φορά τον Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και Υπουργό των Οικονομικών κύριο Λιτζιέ Γεντέας. Παλιός μας γνώρι μα. Τον έχουμε δει πόσες φορές. Αλλά πάντα με μεγάλη επιτυχία στις συζητήσεις μας. Και ήθιστε η απερχόμενη Προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ να ενημερώσει τους ευρωβουλευτές για τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και τις προκλήσεις. δεν είστε απερχόμενοι, αλλά απελθούσα Προεδρία, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως είπαμε ήταν πολύ επιτυχής. Και είμαι πολύ ευτυχής που έστω και με μια μικρή καθυστέρηση έχω την χαρά να σας δώσω την ευκαιρία να μας μιλήσετε για την Προεδρία σας και για τα όσα μας επιφυλάσσει στο μέλλον. DJ, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Σάρων για την πρόταση για την πρόσκληση να έρθω και για την ε, παρουσίαση. Με χαρά βλέπω και πάλι τους ευρωβουλευτές. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν καθήκον ε, βαρύ, ήταν η χαρά να σας συναντώ πάντα συνεδριάσεις και επί της ευκαιρίας σας ε, εύχομαι και ευτυχισμένο το νέο έτος. Έχουμε Ουγγαρία και Πολωνία για τις προεδρίες, τους εύχομαι κάθε επιτυχία, όπως άλλωστε και σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος στην Επιτροπή σας. Δεν θα ήθελα να εξηγήσω περισσότερο, ξέρετε, ότι ήταν δι σκολή η προσπάθεια του συντονισμού με τη Βελική Προεδρία και στη διαδικασία της συναπόφασης ιδιαιτέρως ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τη διαδικασία πάντως, ήθελα να πω ότι από τον Ιούλιο του 2010 στόχος μας ορίστηκε να οργανώσουμε και να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο ε, τα νέα στοιχεία της διαδικασίας συναπόφασης που ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Θεώρησε ότι ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις Αφενό να ξεκινούν οι διαπραγματεύσει αφενός με το Συμβούλιο, αφετέρου με το Κοινοβούλιο, αλλά πάντω ταυτόχρονα ώστε να μην πέσουμε στο αδύνατο εγχείρημα να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Συμβούλιο πρώτα και μετά να περάσει το θέμα στο Κοινοβούλιο ή το αντίστροφο πρώτα να γίνει πρώτα ένα στο Κοινοβούλιο και μετά στο Συμβούλιο. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια ο καθένα εμένει στι δικέ του θέσει και αυτό σημαίνει ότι καθυστερούμε και περνούν μήνε ή και χρόνια ακόμα για να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Γι' αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε ταυτόχρονα και από τι δύο πλευρέ από 1η Ιουλίου. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Είχαμε πρώτο το θέμα της εποπτείας και της νέας αρχιτεκτονικής της εποπτείας. Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε από 1η Ιουλίου, όπως είπα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν ήταν μόνο στόχος της Προεδρίας μας να το, εξασφαλίσουμε αυτό, αλλά... Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω σε ένα Σάρων, αλλά και πολλούς από τους ηγητές σας και τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ διότι σημαντικό ήταν το ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε από πλευράς του Κοινοβουλίου στην αναβολή ορισμένων ψηφοφοριών. Δεν θα επανέλθω, δεν θα ξανανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα είναι πολύ σαφέ ότι ήμασταν στο ίδιο μήκο κύματο, είχαμε το ίδιο όραμα, τη δυνατότητα δηλαδή να διαπραγματευόμαστε και να καταλήξουμε συμφωνία μέχρι το Σεπτέμβριο. Και την ίδια διαδικασία την ξεκινήσαμε και για την οδηγία για το Διεθνέ Ταμείο, που μα επέτρεψε έτσι να προχωρήσουμε σε ένα μέρος τουλάχιστον της νέας νομοθεσίας για, τις, ε, για τους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Και έτσι έχουμε τη νέα αυτή αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι καταφέραμε ομόφωνα στο Συμβούλιο και ευρύτατη, με ευρύτατη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε έγινε και για τις χρηματοπιστωτικές οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, Δυνατότητα, αλλά και για το οδηγία για το Διεθνέ Ουσιαστικό Ταμείο και πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο και για τι λοιπέ ε, οδηγίε που βρίσκονται τώρα εν εξελίξη και που θα ολοκληρώσουν οι επόμενε ε, προεδρίες. Αλλά πάντως πιστεύω τώρα, ότι στις αρχές του 2011, έρχεται η στιγμή για την εφαρμογή αυτού του νέου πακέτου μέτρων, αυτής της νέας αρχιτεκτονικής δηλαδή, και είναι απαραίτητο το ταχύτερο δυνατό να ξεκινήσουμε με τους νέους αρμόδιους και τις νέες αρχές, νέους φορείς για τις αγορές και για τις εταιρείε. Ο Επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ κατέστησε δυνατό το να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σε, με μια προσπάθεια για ένα κατάλογο συγκεκριμένων θεμάτων, ένα shortlist για τις ε, προεδρίες και βέβαια θα οργανώσουμε, όπως ξέρετε, και μια ακρόαση για το κοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο ε, πριν από τον προσδιορισμό και τον, τον προσδορισμό των υποψηφίων και τον διορισμό των νέων προέδρων αυτών των φορέων και των εποπτικών αρχών, γιατί έχουμε αποφασίσει από κοινού ότι η, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να αναλάβει και την προεδρία της νέας αυτής επιτροπής χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, εποπτείας. Ε, αυτά λοιπόν, και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο, αλλά και να αντλήσουμε τα πρώτα διδάγματα όπως άλλωστε κάναμε, της χρηματοπιστωτικής κρίσεως, με τους νέους κανονισμούς, με τις νέες αρχές που θεσπίζονται και ελπίζω, όπως άλλωστε είμαι βέβαιος πως ελπίζει και το, λοιπό, το, το μεγαλύτερο μέρος του Κοινοβουλίου, ε, Ελπίζω λοιπόν ότι χρόνο με το χρόνο θα ενισχύεται η ευρωπαϊκή διάσταση και το ευρωπαϊκό όραμα μέσα στο χρηματοπιστωτικό τομέα θα κρυθεί από το μέλλον αν είναι επιτυχής αυτή η προσέγγιση και αν θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και περισσότερες ακόμη εξουσίες στις νέες αυτές αρχές και ιδίως στην ΕΣΜΑ την Επιτροπή δηλαδή Εποπτεία των Αγορών, γιατί είχε γίνει αυτή η συζήτηση σε σχέση με τους ε, φορείς αξιολόγησης χρηματοπιστωτικής ικανότητα κτλ. Σε μια δεύτερη φάση, επειδή εργαστήκαμε πολύ σε αυτή την περίοδο, να σας πω μερικά λόγια για την διακυβέρνηση. Έγιναν ε, πολλά πράγματα κατά την ε, Βελγική Προεδρία στο Συμβούλιο. Ε, δίπλα στον κύριο Βαν Ρομπόη υπήρξε μία task force η οποία ασχολήθηκε με θέματα διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα το έκανε και η Προεδρία για να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. και θα γίνει μία συζήτηση σχετικά με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Την τελευταία φορά είχαμε πει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ότι οι συγητές θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους και στα τέλη του δευτέρου τριμήνου του 2011 Ελπίζαμε να έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε ούτως ώστε να ξεκινήσει και η συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Αντίστοιχα δηλαδή ότι έγινε με την εποπτεία. Ε, τα κείμενα έχουν παρουσιαστεί από την ε, Κομισιόν, η Task Force έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία φάση εφαρμογής της διακυβέρνησης. Κατά τη Βελγική Προεδρία εμείς μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις... Ε, ε, τώρα για, για το υπόλοιπο των εργασιών μας θα πρέπει να το συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο. Έχουν γίνει συζητήσεις στο Συμβούλιο για τις κυρώσεις και τι είδους κυρώσεις θα πρέπει να, υποβληθ, να επιβληθούν στα κράτη που δεν θα σεβαστούν ή θα γνωρίσουν τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητες. Όλα αυτά όμως είναι καθαρά προπαρασκευαστικά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστεί σχετικά. Για την φορολογία επίσης Εργαστήκαμε ε, κατά την περίοδο της ε, ε, Προεδρίας. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, κυρίως για το θέμα του ΦΠΑ, τεχνικά θέματα. Όμως προχωρήσαμε ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της απάτης σε διοικητικό επίπεδο. Δεν ήταν απαραίτητο να, κυρίως για τις χρηματαγορές να έχουμε ομοφωνία, προσπαθήσαμε να την ε, πετύχουμε αυτή την ομοφωνία για τη φορολόγηση, όμως για τα φορολογικά συστήματα χρειαζόταν ομοφωνία. Παλέψαμε λοιπόν να προωθήσουμε τα ζητήματα που αφορούσαν στην καταπολέμηση της απάτης, διότι όταν καταπολεμάται η απάτη τότε τα κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Υπάρχει όμως ακόμα το θέμα του τραπεζικού συστήματος που το συζητήσαμε πολλές φορές και που θα συνεχίσει να συζητιέται. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν το συζητήσαμε μόνο στο Συμβούλιο, θελήσαμε να το προθίσουμε και σε επίπεδο Διεθνούς Οικονομικού, Οικονομικού Ταμείου και άλλα διεθνή φόρα σχετικά με τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ε, ξεκινήσαμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα πρέπει να μελετήσει όλες τις ε, εφαρμοστικές λεπτομέρειες, τα πρακτικά ζητήματα, δηλαδή ποια θα είναι η φορολογική βάση κλπ. Και ε, υπάρχει όμως η πολιτική βούληση, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε αυτού του είδους ε, την φορολόγηση. Πρόκειται λοιπόν για θέματα στα οποία θέλαμε πραγματικά να προχωρήσουμε. Προσπαθήσαμε κατά την Προεδρία μας να προχωρήσουμε ως προς την ποιότητα των δημοσιοοικονομικών. Όχι απλώς να αναρωτηθούμε αν τα κράτη-μέλη σέβονται τους αριθμητικούς όρους του Μάστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας, δηλαδή έλλειμμα 3%, ε, μικρότερο του 3%, του ΑΕΠ και χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Θελήσαμε να δούμε και την ποιοτική πλευρά, μπορούμε εμείς να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, ας πούμε στην εκπαίδευση, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε μία κοινωνία της γνώσης, μια κοινωνία η οποία γερνάει, ε, αν θα μπορέσουμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε τις συντάξεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε αυτά τα ζητήματα, τα παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα των συνταξιοδοτικών πολιτικών, για την υγεία και για την εκπαίδευση. Δηλαδή θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε τον προϋπολογισμό και ως προς το περιεχόμενό του. Επίσης για τις στατιστικές. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία. Οι στατιστικές δηλαδή να είναι ικανοποιητικές για να μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε τη συζήτηση ακόμη περισσότερο στο τομέα των δημοσίων δαπανών. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για καλύτερη εκπαίδευση οτιδήποτε άλλο αν δεν έχουμε ενιαία στατιστικά στοιχεία ποιοτικά για όλη την Ένωση. Επίσης, πέρα από αυτή την ανάλυση περιεχομένου του προϋπολογισμού, ε, θελήσαμε να προχωρήσουμε και σε μία ανάλυση της εκπροσώπησης των κρατών μελών και της Ένωσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε άλλα φόρα. Θελήσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο για να λάβουμε υπόψη πώς μπορούμε, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε καλύτερα την εκπροσώπηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο G20. Φέτο οι Γάλλοι θα προεδρεύουν του G20. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε μία σύγκληση σε όλα αυτά. Κάποια στιγμή η εκπροσώπηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο G20 εκ μέρους της Ένωσης θα πρέπει να είναι η ίδια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία ε, σταθήκαμε. Δεν θα σας αναφέρω όλους τους εισηγητές και όλους οι εισηγητές που συνάντησα αυτό το εξάμεινο. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής όμως που το συνάντησα, όπως επίσης και οι συνεργάτες μου. Μπορέσαμε να εργαστούμε αποτελεσματικά για τη θετική απόλυξη πολλών κειμένων. Όταν ψηφίζουμε, όταν αποφασίζουμε, είτε στο Κοινοβούλιο είτε στο Συμβούλιο, ε, πάντα έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ένα ποτήρι είτε γεμάτο είτε άδειο. Αν εσείς έχετε το αίσθημα ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο, θα πρέπει να παλέψετε ώστε στην επόμενη Προεδρία το ποτήρι να γεμίσει και να είναι ικανοποιητικό για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε σε αυτό το εξάμεινο και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Ξέρετε ότι εμείς εργαζόμαστε ως τρίο, ε, ξεκινήσαμε τις εργασίες μας υπό Ισπανική Προεδρία και θα συνεχίσουμε στην, κατά την Ουγγρική Προεδρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι οι ομιλητέ μας, οπότε Ζαν Πολ αρχίζουμε με σένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ, Πρόεδρε του ΕΚΟΦΗΝ, επίτιμο πρόεδρο, αλλά είναι ενεργεία παρόλα αυτά. Θα είμαι σύντομος για να έχουν και οι συνάδελφοι χρόνο να παρέμβουν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθέσή μας. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά από πλευράς του ΕΛΚ. Καλό 2011 και καλή επιτυχία. Μας συνηθίσατε σε δυναμικότητα, σε μεγάλες επιτυχίες. Και πάλι εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωσή σας, ε, ε, για τις προσπάθειές σας χωρίς τις οποίες δεν θα είχε τηρηθεί η προθεσμία που είχαμε ορίσει για να καταλήξουμε στις νέες νομικές πράξεις. Σταματώ με τις φιλοφρονήσεις για να σας υπενθυμίσω κάτι και να σας ζητήσω και κάτι άλλο. Δεν ήμουν εγώ εισηγητής και ήθελα να αναφερθώ ε, στην εποπτεία. Όταν μιλήσατε τότε για την εποπτεία στην Ολομέλεια, είπατε ότι πρόκειται για ιστορική καμπή στην Ευρώπη. Δίκιο έχετε ε, και νομίζω ότι κάναμε ένα άλμα όλοι στην Ευρώπη. Και χωρίς να προσθέσω στοιχεία, θα ήθελα να σας μιλήσω για την επιλογή των ατόμων, για τις αρχές. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η επιλογή. Ε, θα ακολουθηθεί η διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι συμβολική η επιλογή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ε, δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών κινδύνων, χωρίς όμως ο πρόεδρος ε, των εποπτικών αρχών να αναγνωρίζεται πέραν κάθε αμφιβολίας από τους υπολείπους. Παρότι δεν παρακολουθούμε όλοι εκ του σε αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα, υπάρχουν εμβλήματα, υπάρχουν σύμβολα που έχουν ιδιαίτερη ισχύ και ελπίζω ότι τα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεχάσουν αυτό που είπατε ότι ο σχεδιασμός της εποπτικής αρχιτεκτονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιστορική σημασία και άρα δεν πρέπει να απολέσουμε τη δυνατότητα που μας δίνεται να εργαζόμεθα πιο αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνω ευχαριστώ σας και πάλι για την ε, συμβολή σας ε, στις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο Ζαν Σωστό αυτό που υπόθηκε για, την, για τις αρχές εποπτείας πρόκειται για μια δοκιμασία, για ένα τεστ. Εμείς δεν ε, ακολουθήσαμε πάντοτε τις θέσεις της Προεδρίας σας, ως σοσιαλιστές, ούτε και τώρα συμφωνούμε 100%, ούτε απαιτείται και να συμφωνούμε 100%, δεν χρειάζεται να ομοφωνούμε όλοι, αλλά να ομονοούμε μάλλον όλοι, αλλά αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι εσείς με πνεύμα ανοιχτό και επικοδομητική προσέγγιση μας βοηθήσατε να προχωρήσουμε περισσότερο, να εξασφαλίσουμε πρόοδο για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό ακριβώς ένα ε, τεστ σοβαρότητας, έλεγχο σοβαρότητας ήταν αυτό το οποίο καταφέραμε για τους πολίτες της Ευρώπης. Και αυτό το οποίο δεν βλέπουν μερικέ φορέ οι πολίτε Ευρώπη είναι ότι μπόρεσαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ευφυα και ε, σύνεση να επιδείξουν και να λάβουν αυτές τις πολύ σοβαρές αποφάσεις για αυτά τα νομοθετήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κανείς έχει προσέγγιση ανοιχτή και επικοδομητική μπορεί να προχωρήσει πολύ και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. ο Διόγκο Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό πρώτα απ' όλα για τις ε, κινήσεις του το τελευταίο εξάμεινο. Επίσης να τον ευχαριστήσω για τις σχέσεις που είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσωπικά θεωρώ ότι μας βοήθησε πολύ για την έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση και τον ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες, για τον τρόπο που συνεργάστηκε με το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα άμεσα να θέσω κάποια ζητήματα. Πρώτον, πώς βλέπετε το μέλλον του ευρώ. Γνωρίζουμε όλοι τι έχει συνέβη. Και σήμερα κάποια δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται ε, σε ισχυρισμού κάποιων σχετικά με την πιθανή χρήση του μηχανισμού στήριξης από πλευρά της Πορτογαλίας. Ε, τι γνωρίζετε εσείς, πώς μπορείτε να τοποθετηθείτε σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα, ειδικότερα, σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την πρόβλεψη που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποχρέωση μείωση των χρεών σε αιτήσια βάση ε, δυνάμει του ε, κανόνα του ενός εικοστού. Επίσης, ποια είναι η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου ε, σχετικά με τις εξαιρέσεις. Μας ενδιαφέρει αυτή η άποψή σας γιατί εγώ ασχολούμαι με το διορθωτικό μηχανισμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρόεδρος, ε, δεν έχουμε χρόνο, οπότε ε, έχουμε ακόμη... Συνεχίζει να ε, διευρύνεται το κατάλογο των ομιλητών. Θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί για να δώσουμε στον Υπουργό τη δυνατότητα να απαντήσει. Ως Βέλγος, όπως και εσείς, ανησυχώ για τη χώρα μου αλλά επίσης ως Βέλγος πρέπει να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα περήφανος για το πώς προείδρευσε το Βέλγιο της Ένωσης. Μπορώ να διαφωνώ στον τομέα σας σε πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι αναλάβατε την Προεδρία σας δυναμικά και με σοβαρότητα. Και φαντάζομαι ότι ε, θα δούμε τη διαφορά με την Ουγγρική Προεδρία. Ελπίζω βέβαια να έχουμε εκπλήξεις, αλλά τέλος πάντων. Για τις εποπτικές αρχές. Μόνο έναν υποψήφιο για ορισμένες περιπτώσεις είχαμε. Αλλά θα ήθελα να σταθώ όμως και σε άλλες υποψηφιότητες οι οποίες αναλύθηκαν. Λοιπόν, για τον πίνακα που πρέπει εμείς να ελέγχουμε, να προσέχουμε. Είπατε στην Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις και το έτανε. Θα ήθελα όμως να ξέρω εσείς τι σκέφτεστε γι' αυτό και τώρα που θα αποκτήσετε και πάλι ελεύθερο χρόνο διότι δεν έχετε πλέον την Προεδρία της Ένωσης και θα παραδώσετε και τη σκητάλη ως ε, αρχηγός του κόμματός σας. Θα σας χαρίσω ένα βιβλιαράκι για τον ελεύθερο χρόνο σας, το οποίο έχει να κάνει με την ε, ανάπτυξη και τις προοπτικές της. Okay, so Ευχαριστώ. Είσαι, είσαι προλάβα να διαβάσω δύο πραγματάκια. Εσεί έχετε τη σειρά. Στου τελευταίου έξι μήνε ουσιαστικά είδαμε δύο πρόεδρες. Τη Βελγική και για πρώτη φορά full time τον μόνιμο πρόεδρο, τον κύριο Φαν Ρόμποϊ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία ή από την έποψή σας πόσο βλέπετε τη σχέση μεταξύ της εναλλασσόμενης προεδρίας και της μόνιμης της μόνιμης Προεδρίας πώς λειτουργήσε, αποτέλεσε πράγματι βήμα προόδου όπως αρχικά είχε προβληθεί η ιδέα ή αποτελεί μόνο μία επιπλέον βαθμίδα της περίπλοκης ούτως ή άλλως, ε, του περίπλοκου ούτως ή άλλως πλέγματος θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος η πλεγματος θεσμων στην ευρωπαικη ενωση ο προεδρος η προεδρος ελληνικου και μετά Τελειώνουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Βελγική Προεδρία για τις ε, προσπάθειές της. Έχει ετοιμάσει πολλούς, πολλά θέματα, έχει προωθήσει πολλούς φακέλους που παραλαμβάνει η Ουγγρική Προεδρία. Βέβαια, η τριανδρία ή τριμερής, ε, το τρίο όπως λέμε, εξασφαλίζει και την συνοχή στη δουλειά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθούμε φυσικά με πολύ ενδιαφέρον τη δουλειά σας, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ε, μετακύληση έμφασης ε, για το πρώτο αλλά και το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς, με την Πολωνική δηλαδή Προεδρία ακόμα. Πολύ συχνά η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη αποτελούν θέμα συζήτησης, αλλά δεν είμαι βεβαία εάν όντως θα την δούμε στην Ευρώπη φέτος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σημειώσω ότι οι επερχόμενες προεδρίες έχουν να κληρονομήσουν αυτές τις μεγάλες δυσκολίε και έχουν και το καθήκον να προσδιορίσουν τους κανόνες εκείνους που θα μας καθοδηγήσουν και πάνω απ' όλα να αγωνιστούν για, το, για τη σταθερότητα του ευρώ. Η Ουγγαρία έχει μια οικονομική πολιτική πολύ καλή και πάνω απ' όλα σύμφωνη με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 σταθεροποιητική δηλαδή πολιτική, με μεθόδους ενδεχομένως ε, που διαφέρουν από κράτος ε, μέλος σε κράτος μέλος, αλλά βλέπουμε ότι οι στόχοι είναι οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είτε πρόκειται για την ε, εταιρική διακυβέρνηση, ε, τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, το νέο ε, δημοσιονομικό προγραμματισμό, την νέα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, τα καθήκοντα που έχει η Ουγγρική Προεδρία, είναι πολύ σημαντικά. Και πιστεύω ότι η καλύτερη προσέγγιση, η πιο επικοδομητική προσέγγιση θα ήταν η συνένεση, το ειλικρινές πνεύμα συνεργασίας και πάνω απ' όλα η αισιοδοξία. Δηλαδή και να βλέπουμε μίσο γεμάτο το ποτήρι και να θεωρούμε ότι μπορούμε να γεμίσουμε αυτό που λείπει από το ποτήρι και να παραδώσουμε ένα γεμάτο τελικά ποτήρι στην Προεδρία της Πολωνίας. Η Ουγγρική Προεδρία είμαι βέβαια ότι θα, θα ήθελε να μελετήσει περαιτέρω αυτά τα καθήκοντα και να συγγραμμιστεί με τις προτάσεις σας. Και, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να εκφράσω ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς τον κύριο Υπουργό για τη δουλειά του αυτό εξάμεινο. Ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο την Προεδρία και κατάφερε να βρει λύσεις εκεί που θεωρούνταν ότι έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο. Και ιδιαίτερα τον ευχαριστώ διότι πάνω απ' όλα αναγνώρισε ότι δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν όλοι στην ίδια θέση και ότι μπορεί να βρεθεί συμβασμός. Πολλά είναι τα κράτη-μέλη και πολλά τα θέματα και οι εκθέσεις που μπόρεσε να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις. Το συγχαίρουμε λοιπόν και τον ευχαριστώ εκ μέρους ε, της Επιτροπής μου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, άξιος ο μισθός σας, μεγάλο το ευχολόγιο που ακούστηκε και τα εγκόμια. θα έχουμε ασφαλώς υπόψη ε, και την ε, προσωπικότητά σα όταν θα έχουμε ενδεχομένως συζητήσουμε το θέμα του Προέδρου του Ίσης και άλλα διάφορα ζητήματα. Δεν θα σας αποχωριστούμε τώρα, έχουμε ένα ποτό οργανώσει εδώ έξω Πάντως περιμένω να μας δώσετε κάποιες τελικές ιδέες. Σας ευχαριστούμε πολύ θετικά τα σχόλιά σας αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να συζητήσουμε με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη. Ε, και προσπαθούμε, ναι, ε, στην Προεδρία μας προσπαθήσαμε να βρούμε μια, ένα συμβιβασμό, αλλά μην ξεχνά τη μακραίωνη παράδοση του Βελγίου για την επίτευξη συμβαστικών λύσεων. Με χαρά συνεργαστήκαμε στους περασμένους μήνες ε, και είμαι σίγουρος ότι τους επόμενους μήνες η Ουγγρική Προεδρία τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει για να ρυθμίσει κάποια δύσκολα και λεπτά ζητήματα. Για... Θα είμαι τώρα, με επικραματικό τρόπο θα σας απαντήσω γιατί δεν έχουμε χρόνο, για την προεδρία των διαφόρων αρχών. Ο στόχος ποιος ήταν να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή εξουσία και αυτονομία ε, και αυτό προέκυψε και από τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να έχουμε ένα σύντομο κατάλογο, ένα short list από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και οι υπόλοιποι να έχουν λάβει άλλε υποψηφιότητε και οι ίδιες οι αρχές να κληθούν να αποφασίσουν χωρί να παρέμβει το Συμβούλιο. Έτσι είπαν κάποιοι και όπω και εσείς ε, ξαφνιάστηκα και εγώ γιατί δεν είχαμε τόσε πολλέ υποψηφιότητε, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όταν ε, έχουμε κάποιον υποψήφιο γυναίκου διστάζουν όλοι οι υπόλοιποι θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια ελπίζω πάντως ότι θα διοριστούν ισχυρέ προσωπικότητε. επικοινωνία επικεφαλή των αρχών για την αρχή συστημικού κινδύνου. Ε, έχετε, έχουμε όλη την τύχη να έχουμε τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, ε, τέλος πάντων δεν θα ήθελα τώρα να τοποθετηθώ. Ούτως ή άλλως γνωρίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ακροάσεις για τους διαφόρους ε, υποψηφίους. Ε, δηλαδή η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι ίδιες εποπτικές αρχές ε, θα ακούσουν τις παρεμβάσεις των υποψηφίων. Οπότε δική σας αρμοδιότητα είναι και δεν το σχολιάσω εγώ για το ευρώ, τώρα την οικονομική διακυβέρνηση και την μακροοικονομική εποπτεία. Και είμαι πεπισμένος ότι χάρη στο ευρώ αντιστεκόμαστε σε αυτήν την ισχυρότατη κρίση που βιώνουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα απαιτούμενα εργαλεία ούτως ώστε να μην έχουμε δυσκολίες τα επόμενα χρόνια με το ευρώ. Είμαι πεπισμένος θα τα καταφέρουμε και εργαζόμαστε και το ίδιο και το Κοινοβούλιο για να έχουμε μηχανισμούς παρέμβασης ε, επαρκώς ισχυρούς ο νέος μηχανισμός ε, φερειπίνη σταθερότητα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα αντικαταστήσει τον, ε, το χρηματοοικονομικό μέσο που είχαμε προβλέψει ήδη από το 2013. Να έχει λοιπόν τα απαιτούμενα μέσα αυτός ο μηχανισμός. Επίσης η ΕΚΤ θα πρέπει να παρεμβαίνει με κάποια άνεση για να εξηγιάνει την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη. αλλά αυτό θα είναι δυνατόν μόνο αν τα κράτη-μέλη όλα δεχτούν την αιρεσιμότητα. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στο μηχανισμό και να αναλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να επανέλθουν ε, σε ισοσκελισμό του προπολογισμού το ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Για την οικονομική διακυβέρνηση, και δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη, αλλά του Συμβουλίου, διαγράφεται μία τάση ε, υπέρ ε, αυτού του στοιχείου, δηλαδή τη ποσοτικοποίηση του δημοσίου χρέου. Ε, αν τώρα θα ακολουθήσουμε τον κανόνα του ενό εικοστού ή όχι δεν ξέρω, αλλά πάντως χρειαζόμαστε ένα ε, σαφώ προσδιορισμένο στόχο και όχι μια γενικόλογη αναφορά για τι κυρώσει τώρα, γιατί υπάρχουν και συζητήσει ε, περί διαδικασίας, αλλά δεν ασχολείται κανεί με την αναγκαιότητα επιβολή κυρώσεων. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα. Μέχρι πού θα φτάσουμε με τι κυρώσει, αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Ε, δηλαδή καταθέσεις με τόκο, χωρίς τόκο, ε, πολιτικές κυρώσεις κάποια μέρα, ε, γιατί μιλήσαμε για αναστολή παραδείγματος χάρη του δικαιώματος ψήφου. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι η καλή λύση, διστάζω ενώπιον μια τέτοια διαδικασία και θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο ενός κράτους μέλους να απολέσει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία. Μήπω είναι υπερβολικό, υπάρχουν άλλα είδη ίσω κυρώσεων και πολιτικών πιέσεων που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και αυτό συνδέεται με τη μακροοικονομική υποπτία και σας είπα προηγουμένως ότι έχουν υποβληθεί εκθέσεις στο Συμβούλιο για τις ε, συντάξει, για την παιδεία, για ε, τον τομέα της υγείας, στη μακροοικονομική εποπτεία. Πιστεύω πάντως ακράδαντα ότι πρέπει πέρα από τα θέματα του ελλείμματος, εξέλιξη του δημοσίου χρέους, ε, τα θέματα ανάπτυξη πληθωρισμού και επιτοκίων, να προσθέσουμε και ζητήματα όπω απασχόληση, ποιότητα των θέσεων απασχόληση, ε, θέματα χρηματοδότησης ε, των δαπανών λόγω της γύρανσης του πληθυσμού ε, πάνε στον τομέα της υγείας και όπως σας είπα έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε τα πετούμενα μέσα για να καταπολεμήσουμε και τις κλιματικές αλλαγές. Όλες αυτές οι παράμετροι θα συνυπολογιστούν. Προφανώς δεν πρέπει να έχουμε υπερπληθώρα παραμέτρων. Η μακροοικονομική εποπτεία χάνει το νόημά της αν δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους που όμως θα είναι επαρκή ώστε να καλύπτεται το περιεχόμενο όλων των δημοσίων δαπανών. Και κλείνοντα ε, θα ήθελα να σα πω πέρα από το ότι ευελπιστώ όπως η Ουγγρική ε, Προεδρία θα μπορέσει να γεμίσει το ποτήρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρομαι στη μεταφορά που κάνατε δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει ποιο ε, θα το αδειάσει όταν το γεμίσουμε αλλά εν πάση περιπτώσει η πολεμική κυβέρνηση μετά την Ουγγρική μπορεί να αποφασίσει να αρχίσει να γεμίζει ένα άλλο ποτήρι και όχι να αδειάσει μόνο το προηγούμενο ποτήρι. Μπορεί να έχουμε πολλά ποτήρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αλλά δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε και το θέμα της ε, λειτουργίας ε, της Προεδρίας. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει, χρειάζεται εδώ να σας υπενθυμίσω πόσο περίπλοκη είναι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ορισμένε φορές. Το ξέρετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Εμείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δύο πράγματα. Πρώτον, όλα όλες οι συναρμόδιες θεσμικές ε, αρχές να συνεργαστούν γύρω από το Eurogroup και το ECOFIN. Πρόεδρος του Eurogroup, έτσι, μόνιμος ε, πρόεδρος ε, του Eurogroup, όπως προβλέπετε, προεδρία του ECOFIN, μόνιμη προεδρία του Συμβούλιου, φυσικά ήμασταν σε άμεση συνεργασία, η προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είδαμε ότι όλα αυτά λειτουργούν εύρυθμα για το, την συνεργασία της Βελικής Προεδρίας με τη μόνιμη προεδρία που επίσης είναι και αληθεύει αυτό προ το παρόν, έτσι. Ε, αυτό προσπαθήσαμε κυρίω να κάνουμε είναι να ε, προβάλλουμε το, στα, το μέγιστο δυνατόν την ε, μόνιμη Προεδρία και να αφήσουμε τη Βελγική Προεδρία να αναλάβει τα συντονιστικά θέματα και ο Βέλγος Πρωθυπουργό νομίζω μπόρεσε να αναλάβει αυτό το συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στι διάφορε συναρμόδιε βελγικές αρχέ και τις συναρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές αλλά όχι να καταλάβει αυτό τον Πρόεδρο που έχει απολέσει πλέον η εκπαιδευτική σε Προεδρία, γιατί έχει αναλυφθεί αυτός ο ίδιος ρόλος από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι υπαρκτή αυτή η εξέλιξη και ίσως ε, ε, αδιαφοροποιούμεθα σε σχέση με προηγούμενε προεδρίες είναι απλούστερο, απλώ να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε δύο διαδοχικού πρωθυπουργού τη ίδια χώρα ε, και του ίδιου πολιτικού προσανατολισμού. Ελπίζω να ακολουθηθεί αυτό το παράδειγμα γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε περιθώριο λιγμών στη μόνιμη προεδρία του Συμβουλίου, τόσο ώστε οι εθνικέ αρχέ να ασχοληθούν με το συντονισμό για τις διάφορες των δράσεων των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου. Ε, και για τα θέματα Συμβουλίου μην ξεχνάτε ότι είναι θέματα ε, του ε, μόνιμου Προέδρου. Ε, Τέλο πάντων, θα συνεχίσει να μετεξελίσσεται ο ρόλο αυτή τη μόνιμη Προεδρία και δεν σα έκρυψα ποτέ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα διαβεβαιώ ότι. Ε, είμαι ευγνώμων. Ποτέ δεν έκρυψα ότι μια ιδρυτική χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω το Βέλγιο έχει τύχη γιατί έχει αξιωματούχου και αρχέ που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά του ευρωπαϊκού μηχανισμού γιατί ε, συμμετέχουν σε αυτού ε, επί σειρά ετών. Μπορέσαμε να συναντηθούμε εδώ στι Βρυξέλλε και ευχαριστώ για όλε τι συναντήσει που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πολύ απλούστερο η Προεδρία να διοργανώνει τι συνεδριάσει στον ίδιο δρόμο έτσι, με την αρμόδια εθνική Καταλαβαίνω πόσο πιο περίπλοκο είναι για άλλε ε, προεδρίες και επίσης είναι ίσως απλούστερο να ε, οργανώνομαστε ανάμεσα σε μια εκπεριτροπή σε Βελγική Προεδρία και μια μόνιμη επίσης Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, έχουμε χαράξει πια το δρόμο και ελπίζω να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Είδου και κλείνω. Ήμουνα επιγραμματικός. Ήταν και μακρά η συζήτηση, αλλά δεν έχω επιλογή. Πάντως, σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία μας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ σε σχέση με προηγούμενες προεδρίες. Ο κύριος Γκόσες ε, ε, μας μίλησε για τον επίτιμο πρόεδρο. Ε, εγώ είχα την τύχη το 2001 και το 2010 να προεδρεύσω του ΕΚΟΦΗΝ και οφείλω να, να ομολογήσω, αν θυμάμαι καλά, ότι το 2001 ε, συναντήθηκα δύο-τρεις φορές μόνο έτσι, με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα το 2010 μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ περισσότερες οι συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές και θεωρώ ότι αυτό από μόνο του συνιστά θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συζητήσαμε πολύ για ποτήρια άδεια, γεμάτα, μισογεμάτα, μισοάδια. Είναι αρκετά λοιπόν αυτά που μας περιμένουν απ' έξω και που είναι πολύ γεμάτα και περιμένουμε να τους δώσουμε την αμέριστη προσοχή μας σε αυτά τα ποτηράκια. Σας βλέπω έξω λοιπόν.